Σας προτείνω να ξεκινήσουμε τις εργασίες μας. Ο πρόεδρος, ο κύριος Λάινεν, θα... δεν είναι παρόν, γι' αυτό θα προεδρεύσω εγώ. Θα, προτείνω, σας πρότεινα να υιοθετήσουμε καταρχήν την ημερήσια διάταξη με τρεις αλλαγές. Στο πέμπτο σημείο, που αφορά το, πρωτόκολλο, το πρόσθετο πρωτόκολλο τη Συμφωνία Συνεργασίας για την Προστασία των Ακτών και των Ιδάτων του Βορειοατλαντικού, Βορειοανατολικού Ατλαντικού από τη ρήπανση. Έκθεση Ροσμπαχ. Αυτό θα το συζητήσουμε στις 2 Δεκεμβρίου το, το πρωί ως τελευταίο σημείο. Σημείο υπαριθμών 17. Δεύτερον, για το σημείο 8 υπάρχει μια ψηφοφορία για τα, επενδυτικά σχέδια σε ενεργειακή υποδομή εντός Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Αναβάλλεται για την επόμενη συνεδρίαση, γιατί τίθεται σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας και γι' αυτό αναβάλλεται αυτό το σημείο. Τελευταίο. Σημείο 14. Για την ασφάλεια του εφοδιασμού της ΕΕ σε φυσικό αέριο. Έκθεση Sonic θα το συζητήσουμε πριν το σημείο 13. Θα αντιστρέψουμε τα σημεία δηλαδή 13 και 14. Το απόγευμα της 1ης Δεκεμβρίου. Με αυτές τις τρεις αλλαγές λοιπόν, συμφωνείτε με την ημερήσια διάταξη. Δεν υπάρχει αντίρρηση. Ευχαριστώ. Για την ε, διερμηνία. Υπάρχει σε όλες ε, τις γλώσσες εκτός από τα λιθουανικά όχι τα λετονικά και τα εστονικά, διορθώνει ο Πρόεδρος. Τρίτο σημείο. Η διάσκεψη που θα γίνει στις 3 Δεκεμβρίου, δηλαδή την ε, ε, Παρασκευή το πρωί στις 10 η ώρα. Όχι, όχι, λάθος, συγγνώμη, λέει η Πρόεδρος, ε, πέμπτη πρωί στις 10 η ώρα. Θα είναι μια διάσκεψη με τον κύριο Πατσάουι που πήρε ε, το βραβείο Νόμπελ για το θέμα της ε, αύξησης θερμοκρασίας του πλανήτη και την ε, επισητιστική πολιτική. Είναι μια ανοιχτή διάσκεψη που θα γίνει μεταξύ 10 η ώρα και 12.30 η ώρα. Ο πρόεδρος, ο κύριος Λάινεν, θα είναι παρόν και όλοι όσοι θέλετε να συμμετάσχετε είσαστε ευπρόσδεκτοι. Τώρα, θα ήθελα να εγκρίνετε τα πρακτικά των συνεδριάσεων 5ης και 6ης Οκτωβρίου, 19ης Οκτωβρίου και 3ης και 5ης, 3ης ε, έως 5ης Νοεμβρίου. Παρατηρήσεις. Σας ευχαριστώ. Το πρώτο ουσιαστικό σημείο της σημερινή μας συνεδρίασης είναι μια ανταλλαγή απόψεων με το Γενικό Διευθυντή, κύριο Φίλιπ Λόβε, που έχω την τιμή να υποδέχομαι σήμερα, είναι δίπλα μου για το θέμα της ε, ανταγωνιστικής συμπεριφοράς στο φαρμακευτικό τομέα. Κύριε Διευθυντά, κύριε Γενικέ μάλλον, αν θέλετε να πάρετε το λόγο και εν συνεχεία θα γίνει συνήθη συζήτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε σήμερα. Θα συζητήσουμε τα πορίσματα και τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προκύπτουν από την έρευνα στο φαρμακευτικό τομέα. Όπως ξέρετε, η πολιτική της Κομισιόν ε, διέπεται από το βασικό στόχο της εξασφάλισης της πρόσβασης σε ασφαλή, καινοτομή και μη ακριβά φάρμακα. Και αυτό είναι μεγάλη πρόκληση. Η νέα ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος Μπαρόζο, αναγνωρίζει τη σημασία αυτής της πρόκλησης και οι Γενικές Διευθύνσεις ε, Επιχειρήσεων και ΣΑΝΚΟ θα συνδράμουν για να αντιμετωπίσουν αυτή την πρόκληση. Και εμείς ε, στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού και εμείς θα συνεισφέρουμε όσο μπορούμε στη συζήτηση για την νομοθετική πρωτοβουλία που έχει αναλάβει η Κομισιόν στον φαρμακευτικό τομέα. Φυσικά, μέσω της εφαρμογής του δικαίου του ανταγωνισμού προσπαθούμε να βοηθήσουμε και εμείς στην υλοποίηση των στόχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως ε, υποστηρίχθηκαν και τροποποιήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να σας εξηγήσω σήμερα τι διακυβεύεται για τους ε, καταναλωτές και ασθενείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιες είναι τα βασικά μελήματα ανταγωνισμού και τι μπορούμε να κάνουμε οι συστάσεις μας ε, εστιάζονται στο, στην ανταγωνιστική σχέση μεταξύ των εταιριών που παράγουν τύπα φάρμακα και γενώσιμα φάρμακα. Ε, αυτά ερευνήσαμε. Όπως ξέρετε, κάθε ασθενής στην Ευρωπαϊκή Ένωση ξοδεύει κατά μέσο όρο περίπου 330 ευρώ το χρόνο για φάρμακα. Και η τάση μάλιστα αυξάνεται οι συνολικές δαπάνες για τα φάρμακα είναι περίπου το 2% του ε, Ευρωπαϊκού ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε όλα τα κράτη-μέλη ε, τα δημόσια ταμεία είναι υποπίεση. Επομένως, οι πολιτικοί σε όλη την Ευρώπη φυσικό είναι να προσπαθούν να κάνουν εξοικονομήσεις για να χρηματοδοτήσουν το σύστημα υγείας. Και φυσικά δεν είναι εύκολο να εξοικονομήσουμε ε, σε ό,τι αφορά τα καινοτόμα φάρμακα όπου οι καινοτομίες αυτές και οι εφευρέσεις είναι σίγουρα πιο ακριβές και γιατί χρειάζονται αρχικές επενδύσεις που κάνουν οι εταιρείε αρχιετύπων φαρμάκων και φυσικά θα πρέπει να ανακτηθούν αυτές οι επενδύσεις που κάνουν εκ των προτέρων. Ε, τα περισσότερα, αν όχι όλα τα κράτη-μέλη, προσπαθούν με ενεργό τρόπο να κάνουν εξοικονομήσεις μέσω των γενώσιμων. Αυτά τα φάρμακα έχουν την ίδια δραστική ουσία με τα αρχέτυπα φάρμακα και γι' αυτό είναι το ίδιο αποτελεσματικά και το ίδιο ασφαλή, αλλά είναι πολύ πιο φθηνά. Και τα φάρμακα αυτά τα γενώσιμα μπορούν να μπουν στην αγορά αυτή τη στιγμή ε, τα αρχέτυπα έχουν χάσει τα δικαιώματα αποκλειστικότητα, ειδικά όταν ε, σταματάνε να ισχύουν τα διπλώματα ευρεσιτεχνία. Στην Ευρώπη, ο ανταγωνισμό μεταξύ των γεννόσιμων φαρμάκων έχουν σκοπό να μειώσουν την τιμή των φαρμάκων, να αυξήσουν την προσπελασιμότητα των φαρμάκων από τους ασθενείς. Παραδείγματο χάρη, τρία χρόνια μετά την εκπνοή του διπλώματο Τεχνίας, η κατανάλωση αυξάνει συνήθως κατά 60%. Και τρίτον, να υπάρχουν κίνητρα για την κοινοτομία. Ε, οι εταιρείε αρχέτυπων θα πρέπει να φέρουν νέα προϊόντα στην αγορά για να υποφεληθούν από τι υψηλέ τιμέ αυτών των νέων φαρμάκων. Α δούμε από πιο κοντά τώρα τι τιμέ των φαρμάκων. Με βάση την έρευνα, ε, τα γενώσιμα μπαίνουν στην αγορά με τιμέ 25% χαμηλότερε από τι προηγούμενε τιμέ των αρχέτυπων. Και είναι 40% ε, πιο φθηνά μετά από δύο χρόνια. Αυτό σημαίνει μεγάλε εξοικονομήσει για τα εθνικά συστήματα υγεία. Επίσης εξετάσαμε αν περισσότερες εξοικονομήσεις θα μπορούσαν να γίνουν μέσω της ε, θέσης ε, στην αγορά των ε, γεννόσιμων και βρήκαμε ότι υπάρχουν σοβαρότερες καθυστερήσεις εισαγωγή στην αγορά των γεννόσιμων με βάση το δείγμα που ερευνήσαμε. Συνήθως χρειάζονται 8 μήνες κατασταθμισμένο μέσο όρο για να μπουν στην αγορά. Και αυτή είναι μάλλον μια συντηρητική εκτίμηση. 8 μήνες μπορεί να σας φαίνεται μικρό χρονικό διάστημα. Αλλά αυτή η καθυστέρηση έχει σημασία. Οι καθυστερήσει έχουν σημασία. Κάθε μέρα καθυστέρηση. μετράει. Γιατί είναι τμήμα του ετήσιου κύκλου εργασιών ενός πολύ πετυχημένου φάρμακου. Ε, συντηρητική είναι η εκτίμηση αυτή. Και αναλύοντας κάποια δείγματα φαρμάκων, οι εξοικονομήσεις από την εισαγωγή των γενώσιμων θα μπορούσαν να είναι 20% μεγαλύτερες εάν η εισαγωγή των φαρμάκων αυτών στην αγορά είχε γίνει νωρίτερα, αμέσως μετά την εκνοή των διπλωμάτων. Ποιοι είναι οι λόγοι καθυστέρησης. Και εδώ θα πρέπει να τονίσω ότι η έρευνά μας, αυτή η τομιακή έρευνα, ε, δεν βασίζεται σε προκατασκευασμένες ιδέες για τους λόγους της καθυστέρησης. Η έρευνα εστίασε σε ένα στοιχείο της καθυστέρησης, που είναι η συμπεριφορά των εταιριών. Και στο βαθμό που συνδέεται με κάποια πτυχή του δικαίου ε, ανταγωνισμού. Δηλαδή, συμπεριφέρεται η εταιρεία με τρόπο κατά του ανταγωνισμού και επομένως θα πρέπει οι αρχές του ανταγωνισμού να την ελέγξουν. Αυτό είναι το θέμα. Παρ' όλα αυτά, φυσικά να γνωρίζουμε ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες δουλεύουν και εργάζονται μέσα σε ένα πολύ ε, περίπλοκο κανονιστικό πλαίσιο και γι' αυτό Πέρα από αυτά που λέμε για την συμπεριφορά των εταιριών, ε, είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε συστάσεις για τις ρυθμίσεις τις ίδιες. Λοιπόν, εξετάζουμε τη συμπεριφορά των εταιριών. Εξετάζοντάς την, βρήκαμε ότι οι εταιρείε αρχιετύπων χρησιμοποιούν διάφορα εργαλεία για να προστατεύσουν τα έσοδά του από τα πετυχημένα τους φάρμακα. Ε, χρησιμοποιώ τη λέξη εργαλεία, όχι γιατί την επινοήσαμε εμείς, αλλά γιατί στην έρευνά μας ε, και στι επιθεωρήσεις μα, όταν ε, κοιτάξαμε τι εταιρείε, αυτές οι ίδιες χρησιμοποιούν αυτή την ορολογία. Ε, εργαλεία, μιλάνε για εργαλεία για να αυξήσουν τα κέρδη τους. Αυτά τα εργαλεία φυσικά ε, υλοποιούν και κάποιου θεμητού στόχου. Με βάση το δίκαιο του ανταγωνισμού ελέγχονται μόνο οι προϋποθέσεις αλλά βεβαίως μπορούν να οδηγήσουν σε άσχημε τάσει. Παραδείγματο χάρη στρατηγικέ για τα διπλώματα ευρεσιτεχνία. Συχνά οι εταιρείε θέλουν να αυξήσουν το, τη διάρκεια και το εύρος ε, της προστασίας, ε, υποβάλλοντας πολλές αιτήσει για το ίδιο φάρμακα. Δηλαδή ε, διπλώματα, δέσμες ε, διπλωμάτων ευρεσιτεχνία. Συχνά ε, τα μεμονωμένα ε, φάρμακα προστατεύονται από 1.300 ε, διπλώματα ευρεσιτεχνία και αιτήσει για διπλώματα σε όλα τα κράτη-μέλη. Έχουμε φακέλου που δείχνουν ότι αυτό είναι ένα από του λόγου που καθυστερούν τα γενώσιμα να μπουν στην αγορά. Και αυτό είναι ιδιαίτερα προβληματικό, γιατί σημαίνει ότι το σύστημα έχει αδυναμίες. Η εφαρμογή των διπλωμάτων ευρεσιτεχνία μέσω των δικαστηρίων φυσικά είναι ένα στεμητό σκοπό. Αλλά από την έρευνα είδαμε ότι η διαφορά ενώπιον του δικαστηρίου γίνεται για να δημιουργήσει εμπόδια στου ανταγωνιστέ και κυρίω στου μικρού ανταγωνιστέ. Οι εταιρείε αρχετύπων θεωρούν τι διαφορέ ενώπιον των δικαστηρίων όχι γιατί έχουν λόγο να το κάνουν, το θεωρούν ότι είναι ε, ένα εργαλείο για να αποτρέψουν τους ανταγωνιστές. Με βάση τα πορίσματά μας, οι εταιρείε ε, γενοσύμων αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα. Και μια διαφορά ενώπιον δικαστηρίου ε, χρειάζεται να διεκπεριωθεί μέσα στα δικαστήρια 2,8 χρόνια. Αν λάβετε υπόψη σας το κόστος της καθυστέρησης που σας είχα πει προηγουμένως, καταλαβαίνετε τι επιπτώσεις έχει αυτό. Ε, η έρευνα λέει ότι μεταξύ του 2000 και του 2007 ή Ιούνιο 2008, οι εταιρείε γενώσιμων και αρχετύπων είχαν περίπου 200 ε, τέτοιες διαφορές. Οι μισές από αυτές ε, περιόριζαν με κάποιον τρόπο την εισαγωγή γενώσιμων στην αγορά. Και ένα σημαντικό ποσοστό σημαίνει, ε, οδήγησε μάλλον και σε μεταφορά ενός ποσού, μια πληρωμή δηλαδή, από τις εταιρείες αρχετύπων στις εταιρείες γενοσύμων. Είχαμε επίσης και 200 εκατομμύρια ευρώ σε άμεσες πληρωμές. Αυτά τα ποσά τα εξέτασαν και στο Αμερικανικό Κογκρέσο, τα αντίστοιχα Αμερικανικά ποσά, ε, το, τις, ε, τους όρους μέσα στους οποίους γίνονται πληρωμές για τις καθυστερήσεις. Και το βάρος της απόδειξης είναι στην εταιρεία η οποία πρέπει να δείξει ότι δεν πληρώνει λεφτά οι εταιρείε αρχιετύπων δηλαδή, δεν πληρώνουν λεφτά απλώ και μόνο για να καθυστερήσουν του ανταγωνιστέ. Επομένω, φέρουν το βάρο τη απόδειξη. Επίση, οι εταιρείε αρχιετύπων συχνά παρεμβαίνουν πριν από τι εθνικέ αρχέ που χορηγούν την έκρηση αδειοδότηση. Και λένε ότι τα γενώσιμα φάρμακα, έτσι ισχυρίζονται, είναι λιγότερο ασφαλή, λιγότερο αποτελεσματικά, κατώτερης ποιότητας ή παραβιάζουν τα δικαιώματα που απορρέουν από τα διπλώματα βερσιτεχνία των αρχιετύπων. Ε, με αυτόν τον τρόπο ε, καθυστερούν ακόμα περαιτέρω οι διαδικασίε κατά τέσσερι μήνε. Και συχνά επίση αμφισβητούν ε, τις αποφάσεις των αρχών που χορηγούν την άδεια ε, εμπορίας. Ε, όμως δικαιώνονται μόνο σε ποσοστό 1 έω 2%. Εμείς αυτή την προσπάθεια λοιπόν που κάνουμε για να ελέγξουμε δεν είμαστε οι μόνοι και άλλες αντίστοιχες αρχές κάνουν το ίδιο. Σε διαβουλεύσεις με τους συναδέλφους μας είδαμε ε, τρει τομεί όπου θα έπρεπε να γίνει κάποια μεταρρύθμιση στο κανονιστικό πλαίσιο. Λέγοντα αυτό, δεν θεωρώ ότι το σώμα όλων των νομοθετικών σχετικών προτάσεων που έχουν γίνει, που έχουν συζητηθεί ε, με το Κοινοβούλιο, ε, δεν είναι σημαντικό. Ε, η έγκριση της αγοράς, ε, τα, τιμολόγια, η ασφαλιστική κάλυψη, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για την εφαρμογή του δικαίου. Έχουμε ξεκινήσει ε, μία διερεύνηση των ε, συμφωνιών ε, διευθέτησης γύρω από τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Και θα εξακολουθήσουμε να παρακολουθούμε αυτές τις συμφωνίες, ιδίως αυτές που περιορίζουν την εισαγωγή των γενώσιμων στην αγορά ή που συνεπιφέρουν μία πληρωμή από τις εταιρείε αρχετύπων στις εταιρείε γεννόσιμων. Αλλά αυτά δεν αρκούν. Γι' αυτό λοιπόν Κάναμε και άλλες συστάσεις πολιτικής στην τελική έκθεση. Να σας πω ποια θεωρώ ότι είναι τα βασικά στοιχεία. Πρώτα πρώτα, επιβεβαιώνουμε ότι χρειάζεται να υπάρχουν κάποιες ευρεσιτεχνίες και να υπάρχει και κάποιο σύστημα για την ένδικη επίλυση των διαφόρων για αυτέ τις ευρεσιτεχνίες. Επίσης θα πρέπει να ε, κάνουμε πιο έντονε προσπάθειε ώστε να υπάρχει ασφαλή δικαίωση, διότι όλοι στον κλάδο επιβεβαιώνουν ότι χρειάζεται να γίνει κάτι τέτοιο και αυτό προκύπτει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση του Δημήτρου Ανταγωνισμού ότι επίση 11% αυτών των υποθέσεων σε διάφορα δικαστήρια διαφόρων κρατών μελών Μα είπαν ότι έχουμε αντιφατικές αποφάσεις σε διάφορες υποθέσεις. Επίση είπαμε ότι το ισχύον σύστημα είναι σχετικά πολύ για όλου. ή τέλος πάντων ε, είναι πάρα πολύ συμφέρον για τους ε, δικηγόρους, γιατί έχουμε 420 εκατομμύρια ευρώ ε, που δίνονται σε δικηγόρους για τα έξοδα αυτών των, αυτών των διαφωνών ενώπιον των δικαστηρίων και προέκυψαν αυτά από αυτή μα την έρευνα. Τώρα, αυτή η άδεια θέση σε εμπορία, σύμφωνα με τα όσα ερευνήσαμε, απέδειξαν ότι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ε, ε, εφαρμόζεται. Όμω θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη συνεργασία μεταξύ των αρχών και έτσι να αναβαθμιστούν οι δυνατότητέ του για να προστατευτούν τα συμφέροντα όλων, κυρίως εναντί αυτών που δεν είναι και τόσο ευαίσθητοι στα δικαιώματα των καταναλωτών. Επίσης, καλέσαμε τα κράτη-μέλη να σκεφτούν κατά πόσον θα πρέπει να υπάρχει κάποιο αυτόματο σύστημα για τα γενώσιμα και για κάποια αρχέτυπα προϊόντα και προσπαθήσαμε να εξετάσουμε αναλυτικά το Ολλανδικό μοντέλο. Επίσης θα πρέπει με την αντίστοιχη πολιτική να διευκολυνθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των γενώσιμων και εδώ ασπαστήκαμε το Ολλανδικό σύστημα. Δηλαδή ο γιατρός να μην ε, συνταγογραφεί το πιο... να μην ένα συγκεκριμένο προϊόν αλλά να συνιστά μια ουσία και ο φαρμακοποιός να δίνει το πιο φτηνό. Και με αυτό σχετίζεται και μια οδηγία παλιότερη του 89. Εδώ σταματώ γιατί φαντάζομαι ότι θα έχουν ένα σωρό ερωτήσει ε, τα, μέλη, οι βουλευτέ. Πάντως ελπίζω ότι σα ε, έδωσε μια ιδέα για το περί τίνο πρόκειται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Γενικέ για όλα όσα μας εξηγήσατε. Οπότε τώρα μπορεί να ξεκινήσει μια πλούσια συζήτηση και προβληματισμός. Και έχει δει το λόγο η κυρία Ροτ Μπέρεντ. Σας ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε. Κυρία Λόου, σας ευχαριστώ. Πάρα πολύ προσεκτικά ε, διάβασα την έκθεση και άκουσα αυτό το οποίο μας είπατε. Για πετε μας ακριβώς ε, αυτή η έκθεση Για ποιο λόγο ξεκίνησε, για, τι, κίνητρο είχε. Μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ φορτισμένη ε, πολιτικά. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο μου φαίνεται παράδοξο το ότι προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λέμε εδώ για τα γεννόσημα, κάποιες καταγγελίες, κάποια παράπονα. Όλα αυτά τα λέει εδώ ο κλάδος φαρμακοβιομηχανίας, όμως στον πραγματικό κόσμο ισχύουν αυτά. Στην εισήγησή σας κύριε Λό είπατε ότι το πιο σημαντικό όσον αφορά τα φάρμακα είναι να έχουμε εγγυήσεις ότι οι ασθενείς μπορούν να βρίσκουν καινούργια φάρμακα, μοντέρνα φάρμακα και ασφαλή. Φάρμακα αποτελεσματικά. Μέχρι εδώ καλά. Μετά όμως μας μιλήσατε μόνο για χρήμα, μόνο για τις τιμές. Δεν καταλαβαίνω επομένω πώ είναι εδώ να έχουμε μια τέτοια έρευνα σε αυτό τον κλάδο που να, να μην τον, τονίζει την καινοτομία, να μην ε, θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ βασικό να υπάρχει έρευνα, να μην έχουμε έτσι μια προσθεμένη αξία στα προϊόντα του κλάδου. Και μιλώ φυσικά για τη βιομηχανία των γενώσιμων και από την άλλη μεριά των γιατί δεν είναι το ίδιο. Καφέ Αυτό επομένω εδώ χρειαζόμαστε. Έτσι. Χρειάζεται να υπάρχει έρευνα στον κλάδο. Και κατόπιν ασχολούμαστε με την τιμολογιακή πολιτική. Και εσείς λοιπόν το μόνο που κάνατε ήταν να μιλήσετε πολύ υπερβολικά για τις τιμές. Βεβαίως και είναι πάρα πολύ σημαντικά το Και στην Γερμανία το ίδιο ισχύει. Όμως, να σας πω κάποια συγκεκριμένα σημεία για την πρόσβαση, η προσβασιμότητα σε αυτά τα φάρμακα. Εντάξει, τα έχουμε. Όποιος θέλει πάει και τα αγοράζει. Το θέμα είναι πόσο πρέπει να πληρώσει. Ε, τι θέλετε να πείτε, ότι όταν έχουμε γενώσιμα είναι πιο εύκολη πρόσβαση. Όμω από την μεριά είπατε ότι έχουμε σημαντικέ καθυστερήσει στην προμήθεια. Οπότε ρωτιέται κανεί, τι κανόνε διέπουν την παραγωγή και διάθεση των φαρμάκων και θέση εμπορία. Και βλέπω εδώ πέρα στη σελίδα 23, στη σελίδα 23 μα λέτε ξεκάθαρα ότι από το 2004 άλλαξε άρδινη κατάσταση και από το 2013 πρόκειται να έχουμε αυτά αποτελέσματα. Πάντοτε συμφωνώ μαζί σας στο σημείο που αναφέρετε ότι είναι δυνατόν να έχουμε εξοικονόμηση δαπανών για το δημόσιο εάν έχουμε περισσότερα γενώσιμα. Δεν είχε κάτι τέτοιο. Δεν μας λέει η έκθεση. Ποιος είναι ο ρόλος της φαρμακοβιομηχανίας όταν ε, ασχολείται και επενδύει σε έρευνα και ανάπτυξη. Αν κάποιο επικεντρώνει προσοχή του μόνο στα ε, γενώσιμα, τι κάνει. Αυτό το οποίο κάνει είναι ότι έχει ήδη αντιγράψει κάποιο αρχέτυπο, το οποίο προϋπήρξε. Άρα προς, προς, προσοχή, να μην και με τα χλωρά μαζί με τα ξερά. Θα πρέπει να είμαστε δίκαιοι σωστή και κυρίως αυστηρή με την φαρμακοβιομηχανία, γιατί υπάρχει και κάποιο καθήκον ηθικό και οικονομικό που έχουν. Πουθενά στην έρευνα δεν μας λέτε τίποτα για τον ε, ανταγωνισμό, δεν μας λέτε για κάποιες παρανομίες. Δηλαδή είναι κάπω ουδέτερη, κάπω απονευρωμένη αυτή η εκθέση. Τι μα λέτε για εργαλεία, μέσα, πολιτική. Ε, καλά, ο καθένα έχει τι μεθόδου του για να μπορεί να αντιμετωπίσει ένα συγκεκριμένο θέμα. Δεν βλέπω τίποτα το αθέμητο σε αυτό. Όλοι μέσα στην νομιμότητα κινούμεθα. Όμω, από την άλλη μεριά, έχουμε κάποια θέματα με τι ευρεσιτεχνίε. Και είπαμε ότι θέλουμε εδώ να ισχύσει όσο είναι πιο ενιαία διαδικασία. Τελευταία μου τώρα παρατήρηση, Πρόεδρε. Αυτή η ενισχυμένη συνεργασία. Εξοικονομούν χρήματα οι υπηρεσίες και αρχές όταν συμφωνήσουν με την καταχώρηση στο Μητρό των Φαρμάκων στη χώρα τους κάποιου φάρμακο. Βέβαια θα πρέπει αυτό το φάρμακο να είναι διαθέσιμο στα φαρμακεία. Γίνεται κάτι τέτοιο. Εγώ θα προτιμούσα να είναι τα πράγματα λιγότερο άναρχα, διότι κάποιοι πρεσβεύουν ενιαίο σύστημα, όπως κάποια κράτη-μέλη, με το οποίο βέβαια δεν είναι σύμφωνες οι φαρμακοβιομηχανίες. Χρειάζεται επαγρύπνηση, χρειάζεται υποπτία, να ξέρουμε τι γίνεται με τις παρενέργειες του κάθε φάρμακο. Και η ΕΜΕΑ, η υπηρεσία του Λονδίνου και η Κομισιόν να προσέξουν περισσότερο τι λένε. Η Σάγκο κάτι θα πρέπει να κάνει γι' αυτό και όχι η φρονοβιομηχανία γιατί αλλιώς θα αλλάξει ο αλλιώ τα ρούχα, θα τα βάλει αλλιώ και έτσι τι δεν θα ωφεληθεί κανένα στην Ευρώπη, παρά μόνο η φαρμακοβιομηχανία. Είναι κάπω συντεχνιακή η έκθεση και θα πρέπει αυτό να μην, να μην συνεχιστεί. Οπότε μην μη, με, μη με παρεξηγείτε, γιατί κάπω παρασύρθηκα και ήμουν συναισθηματικά φορτισμένη τώρα που σα μίλησα. Η πρόεδρο. Ε, Ευχαριστώ, κύριε Γενικέ. Θα θέλετε να απαντήσετε. Δεν έγιναν πάρα πολλέ παρεμβάσει. Νομίζω ότι είναι πιο ενδιαφέρον να ακούσουμε λίγε ερωτήσει και αμέσω μετά την απάντηση. Ευχαριστώ κυρία Ροτ Μπέρεντ για τις παρατηρήσει σας. Η παρέμβασή μας με την τομιακή έρευνα, ε, και νομίζω να το είπα και στην αρχή, δεν είχε σαν σκοπό να επιλύσουμε όλα τα προβλήματα του τομέα της υγείας και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τη συμπεριφορά των κρατών μελών. Χωρίς τη δική σας παρέμβαση, χωρίς την παρέμβαση της Επιτροπής, χωρίς την παρέμβαση των ρυθμιστικών αρχών και ελπίζω ότι δεν το ισχυριζόμαστε αυτό στην έκθεσή μας. Δεν νομίζω ότι το λέει πουθενά η έκθεση. Σε ό,τι αφορά την προστασία των δραστηριοτήτων εκείνων που προωθούν την καινοτομία, νομίζω και αυτό το είπα ξεκάθαρα στην αρχή, οτιδήποτε και να κάνουμε στο το δίκαιο του ανταγωνισμού, θα πρέπει να το σεβαστούμε αυτό και να το προωθήσουμε, γιατί ο ανταγωνισμός υπάρχει μόνο όταν οι άνθρωποι που προωθούν την καινοτομία αμείβονται. Τούτου λεχθέντος νομίζω ότι όχι μόνο από την έκθεσή μας, αλλά από πολλές εκθέσεις θα βλέπετε ότι οι νέες καινοτομίε. Ε, οι νέες εφευρέσεις δεν είναι πολλές, είναι λιγότερες. Και όχι αυτό δεν οφείλεται στην Κομισιόν, ούτε καν στην τομιακή μας έρευνα. Οφείλεται σε κάποιο βαθμό δυσκολιών προφανώς που αντιμετωπίζουν οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες που έχουν ακόμα, ακόμα και σήμερα έχουν τεράστια, τεράστιο προϋπολογισμό αλλά αντιμετωπίζουν προβλήματα παρόλα αυτά. Φαντάζομαι ότι καταλαβαίνετε ότι ο βαθμός ε, της κοινοτομίας δεν μειώθηκε λόγω των ε, επιθεωρήσεών μας και τη ερευνά μας. Εμείς εστιάζουμε στην πτυχή της ε, παραγωγής των φαρμάκων και της θέσης στην εμπορία τους που ενδεχομένως να έχουν αρνητικές επιπτώσεις. Το ξαναλέω ακόμα μια φορά. Δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε μια πλήρη τομεακή έρευνα όλων των πτυχών θετικών και αρνητικών του κλάδου. Απλώς να εξετάσουμε, όπως και γίνεται στην έρευνα, το δυναμικό που υπάρχει για αντι, ανταγωνιστική συμπεριφορά ε, σε αυτόν τον τομέα ε, μεταξύ των εταιριών που παράγουν αρχέτυπα και γενώσιμα φάρμακα. Και δεν αποκλείεται ε, κατά την εφαρμογή του νόμου να υπάρχουν και προβλήματα στη συμπεριφορά των εταιριών γενοσύμων. Και εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να το... Έχουμε κάποιους λόγους για να θέλουμε να τις ε, διερευνήσουμε και αυτές τις εταιρείε. Τρίτον, αν είχαμε πει οτιδήποτε για μια συγκεκριμένη εταιρεία ή ομίλους εταιρεών σε αυτή την έκθεση, το οποίο θα ήταν ισχυρισμο εσείς θα ήσασταν οι πρώτοι που θα μας λέγατε ότι είμαστε... Έχουμε λάθος στάση γιατί είμαστε παράνομοι στη συμπεριφορά μας. Ήμασταν πολύ προσεκτικοί λοιπόν και σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να διατυπώσουμε ισχυρισμού, ε, οι οποίες δημιουργούν πρόβλημα στα δικαιώματα των εταιριών ε, αρχετύπων ή γενοσύμων φαρμάκων. Και δεν θέλουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε προβλήματα στα δικαιώματα των εταιριών. Γι' αυτό η έκθεσή μας είναι πιο βαρέτη βέβαια, αναγκαστικά και περιορίζεται σε γενικόλογα σχόλια. Σε ό,τι αφορά το δίκαιο των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. συμφωνώ με τους βουλευτές που είπαν ότι πρέπει να κάνουμε πολλά ακόμη, ούτω ώστε το σύστημα των διπλωμάτων στην Ευρώπη να γίνει πιο αποτελεσματικό και να προωθεί την ε, καινοτομία και τον καταναλωτή τελικά. Πιστεύουμε, πιστεύουμε ότι το Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας έχει ανεβάσει τον πύχη, ε, ειδικά σε ό,τι αφορά τα αδύναμα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Αλλά παρόλα αυτά πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα σε αυτό το τομέα. Και θα τελειώσω με, αυτό το στοιχείο απαντώντας στην ε, κυρία Ροτ Μπέρεντ. Ναι, η νέα Κομισιόν θα πρέπει να κοιτάξει προσεκτικά και να εξασφαλίσει ότι οι πολιτικές της οδηγούν σε συγκεκριμένα και θετικά αποτελέσματα και όχι μόνο σε ρητορίες και φαντασιολογίες. Και θα πρέπει οι υπηρεσίες της Κομισιόν ε, με συνδυασμένο τρόπο να το επιτύχουν αυτό. Ε, και αν αυτό μπορεί, σε, αυτό σε αυτή την προσπάθεια η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού ε, βοηθήσει, τόσο το καλύτερο. Σας ευχαριστώ κύριε Γενικέ. Και τώρα η κυρία Κατρίν Σουλιέ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μία ερώτηση η οποία συνδέεται με την προηγούμενη παρέμβαση. Κύριε Γενικέ, αναφερθήκατε στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα οποία στην Ευρώπη ε, δίδονται σε εθνική βάση και όπως είπατε από το Ευρωπαϊκό Γραφείο ε, Διπλωμάτων που στην πραγματικότητα είναι ένα άθροισμα εθνικών διπλωμάτων ευρυστεχνίας και αυτά υπόκειται στους εθνικούς κανόνες των ε, συμβαλωμένων κρατών και τα εθνικά δικαστήρια είναι αυτά τα οποία που αποφαίνονται σε περίπτωση διαφοράς. Επι, επι, μιλήσατε για ε, ενστάσεις, για προσφυγές. Πότε θα αποκτήσουμε κύριε Γενικέ, ένα πραγματικό ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνία. Απλή είναι η ερώτησή μου. Θα ήθελα να μου απαντήσετε. Μπράβο, λέει η πρόεδρο. Ε, η ερώτηση ήταν απλή τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν η απάντηση ήταν απλή, αλλά η ερώτηση ήταν πάντω απλή. Είμαι ένα ταπεινός γενικός διευθυντής. Ε, και θα πρέπει να, έχω μια, να σας δώσω μια ταπεινόφρονα απάντηση. Είπατε, ότι επειδή δεν υπάρχει ευρωπαϊκό διπλωματικό, ε, ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, έχουμε πολλές ε, απώλειες ε, κονδυλίων. Απώλειες και στην πολιτική μας. Και ελπίζω ο νέος Επίτροπος, όχι μόνο υγείας, αλλά και καινοτομία και έρευνας, αλλά και ανταγωνισμού, ο νέος Επίτροπος Ανταγωνισμού δηλαδή, όλοι αυτοί οι επίτροποι μαζί θα κάνουν συνδυασμένες προσπάθειες για να πείσουν τα κράτη-μέλη και εσά βεβαίω για τη χρησιμότητα ενός ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Ευχαριστώ. Κυρία Άντερ, έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Γενική Διευθυντά. Δεν μπορώ να πω ότι υποστηρίζω τις εταιρείες αρχετύπων φαρμάκων, ούτε τις εταιρείες γενοσύμων. Δεν είμαι με το μέρος ούτε του ενός ούτε του άλλου. Θα ήθελα να σας πω όμως, να σας πω κάτι από τη σκοπιά του ασθενούς ή του δυνητικού ασθενούς. Θέλω να σας πω το εξής. Η έκθεσή σας όσο σωστά διατυπωμένη και προσεκτικά διατυπωμένη κι αν είναι, χρησιμοποιεί στερεότυπα για να περιγράψει το πώς και το πότε οι εταιρείε αρχετύπων χρησιμοποιούν αθέμητες πρακτικές εμπορίας και ανταγωνισμού. δίδοντας παραπλανητικές πληροφορίες στον ασθενή, είτε μέχρι φυλα... μέσω φυλαδίων, είτε μέσω διαφημίσεων στην ε, τηλεόραση, για τα γενώσιμα φάρμακα. Δίδονται λοιπόν λανθασμένες πληροφορίες στους ασθενείς για τα γενώσιμα. Εδώ τίθεται το θέμα του αθέμητου ανταγωνισμού και των αθέμητων εμπορικών πρακτικών κάτι που σαφώς παραβιάζει τα δικαιώματα των ασθενών. Γιατί αν εγώ ως ασθενής ε, λάβω εσφαλμένες ή παραπλανητικές πληροφορίες για ένα φάρμακο, φυσικά θα έχω μία βεβαιότητα για το αν θα πρέπει να χρησιμοποιήσω αυτό το φάρμακο ή όχι. Επομένως το ερώτημά μου είναι, στις περιπτώσεις που αναφέρατε εσείς. πολύ προσεκτικά ε, μιλήσατε για αυτές, αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω. Ποια είναι η πρόταση του συντάκτη της έκθεσης. για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη συμπεριφορά. Αυτή τη συμπεριφορά αυτών των ε, εταιριών. Είναι εθνική αρμοδιότητα η αντιμετώπιση αυτή ή η Κομισιόν σκοπεύει να κυρώσει, να ε, τιμωρήσει αυτές τις συμπεριφορές. Σκοπεύει να κάνει κάτι η Κομισιόν. Λόγω. Νομίζω ότι πέρα υπάρχει μια ποικιλία διαφορετικών ε, στάσεων και συμπεριφορών που θα πρέπει να ερευνηθούν και να διερευνηθούν είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εάν πρόκειται για κάποια στάση που αφορά όλες τις ε, αγορές ή καμιά φορά θα πρέπει αυτό να γίνει σε εθνικό επίπεδο, από το οποίο και ξεκινώ. Μια αγορά σε εθνικό επίπεδο. Ίσως ε, πρόκειται για κάποιες ε, αθέμητες πρακτικές άσκηση εμπορίας όπως παραπλανητική διαφήμιση εκ μέρους του κλάδου ή του τομέα των γενώσιμων ή παραπλανητική διαφήμιση από τον κλάδο των αρχιετύπων. Όμως αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, α πούμε, όταν λέει κάποιο ε, τον αρχέτυπο, μην το χρησιμοποιείτε αυτό, γιατί δεν είναι τόσο ασφαλέ όσο το δικό μα που είναι το αυθεντικό. Ε, τότε σε αυτή την περίπτωση οι αρχέ υπεύθυνε για την έγκριση θα πρέπει να επέμβουν και ε, επέμβουν κατά αυτό που διατυπώνει του ισχυρισμού. Όμω, εάν κάποιο κατασκευαστή ισχυρίζεται ότι ένα φάρμακο θα πρέπει θα, θα, ότι το είναι πιο φτηνό χωρίς να, να το τεκμηριώνει, τότε και εδώ θα πρέπει κάποιος, ε, κάποια εθνική αρχή θα πρέπει να προσφύγει εναντίον ε, αυτού που διευθύνει τους ισχυρισμού επί τη βάση εμπορικής νομοθεσίας. Επίσης τώρα παρακάτω έχουμε κάποιου είδους συμπεριφορές οι οποίες εμείς ως αρχή επί του ανταγωνισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και οι συνάδελφοι σε εθνικό επίπεδο πρέπει να εξετάσουν. Όταν δηλαδή προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια, κάποια, κάποια εισαγωγή φαρμακού τόσο ώστε να μην εισάγονται γενώσιμα. Ή όταν υπάρχουν κάποιε συμφωνίε μεταξύ του κλάδου των γενώσιμων και των χετύπων ει των καταναλωτών. Και είναι εδώ να γίνει και μεταξύ ε, αυτών των γενώσιμων τους ώστε να έχουμε πάγωμα των τιμών ακόμα και όταν έχουμε κάποια ευρεσιτεχνία η οποία έχει εκπνεύσει, έχει, έχει, έχει, έχει, έχει εγκαταληφθεί έχει απεμποληθεί από τον αρχέτυπο. Οπομένω, κάποιε από αυτέ τι συμπεριφορέ είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν από την Κομισιόν ω αρχή του ανταγωνισμού. Άλλε συμπεριφορέ προσυδειάζουν σε συγκεκριμένε χώρε. Οπότε και το πιο σωστό είναι η Εθνική Αρχή Ανταγωνισμού να τα αντιμετωπίσει. Και αυτό και κάνουν τώρα. Σας παραλαμβάνω ότι εμείς δεν προσπαθούμε να κηρύξουμε την αρχή της συνωμοσία. να ξεκινήσει μια πλημμύρα καταγγελιών κλπ. Δηλαδή να λέμε ότι η διαφήμιση είναι, είναι, είναι, είναι παραβίαση εμπορικής νομοθεσίας ε, κλπ. Ή να καταλήξουμε σε κάποιους περιορισμού κάποιων ε, δραστηριοτήτων ε, κάποιων ανταγωνιστών. σε περίπτωση που θα έπρεπε να γίνει καλύτερη διάκριση μεταξύ του προϊόντος του μεν από τα προϊόντα των υπολείπων. Πολλές φορές επίσης θα πρέπει να εξεταστούν κάποιες περιπτώσεις όπου συντρέχει λόγος στη δύναμη της ε, νομοθεσίας του ανταγωνισμού Πολλές φορές έχουμε κάποιες ε, επιλήψεις με συμφωνίες, ε, συμφωνίες που περιθωριοποιούν, ξερούν κάποιους, αυτό μπορεί να ισχύει και από πλευρά εθνικών αρχών, μεταξύ χωρών. πάση σε κάθε εθνική νομοθεσία θα πρέπει να εξετάζει πώ αποφεύγεται η παραπληροφόρηση του καταναλωτή και η παραπλανητική διαφήμιση. Και αυτά είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν από το εθνικό δίκαιο. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο τώρα. Ενδεχομένω χωρί περίπτωση προσφυγή, περίπτωση τον να επικαλεστεί κανείς το ε, κοινωτικό δίκαιο και να προσπαθήσει να το εφαρμόσει σε περίπτωση κάποιας ε, πραγματικής διαφήμισης σε εθνικό επίπεδο. Τι λέει. Ναι, κύριε Σλούτο. Thank you for coming here. Contrary to many of my friends... Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Με μεγάλη χαρά έχουμε την έκθεσή σας, διότι πολλά μπορούμε να κερδίσουμε και να εξοικονομήσουμε αν λειτουργήσει ο νόμος όπως το χεύγουμε. Και θα πρέπει εδώ να λάβουμε υπόψη το διάστημα των 20 ε, ακριβώς ε, ετών. Γιατί μόνο σε, κάποια, σε κάποιες λίγες περιπτώσεις όταν υπάρχει ε, υπόθε, περίπτωση να εφεσιβάλλουν τότε μπορεί αυτό να ρυθμίζεται με βάση αυτές τις διατάξεις. Σε σχέση με τις, ε, ε τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας ε, βαίνει καλώς η ρύθμιση, όμως ε, ένα πιο ευαίσθητο θέμα δεν το θίγεται και αυτό θα ήθελα να κάνω. Δύο τμήματα, το ίδιο το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας πρώτα, όσον αφορά την καινοτομία. Αν μπορεί κανείς 100 ευρεσιτεχνίες χρειάζονται για να μπορέσει να καλυφθεί και να κατοχυρωθεί ένα φάρμακο αυτά τα 100 διπλώματα έβρεση τεχνίας ε, με αυτόν τον τρόπο μπορούν να δικαιολογήσουν την ύπαρξή τους και όταν έχουμε με ένα φάρμακο δεύτερης γενεάς και χρησιμοποιείται μια διαδικασία για να σταματήσουν τα γενόσχημα που ε, αντιγράφουν τα αρχέτυπα. Όταν έχουμε ένα φάρμακο δεύτερης γενεάς, τι γίνεται. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ε, όσον αφορά την καινοτομία δεν επακούσε είναι ένα τεράστιο πρόβλημα διότι στραγγαλίζει τον ανταγωνισμό. Αν μόνο όταν υπάρχει μια ε, σοβαρή καινοτομία χορηγείται ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Αυτό Ούτω έχει πρέπει να προσαρμόζεται όταν χορηγείται ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνία. Έχω την εντύπωση ότι πολλέ φορέ λειτουργούν τα πράγματα διαφορετικά. Και οι ομάδε ευρεσιτεχνιών. Καμιά φορά χρειάζεται μια συγκεκριμένη διαδικασία για να μπορεί κανείς να παράξει ένα φάρμακο. Και μέσα από ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που καλύπτει, ας το πω έτσι, μια τέτοια διαδικασία, μπορούμε να αποφύγουμε ε, οποιαδήποτε προσβολή. Έχετε εσείς ε, δει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια τέτοια διαδικασία σε σχέση με ένα παλαιό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Δεν υπάρχει ποτέ μια περίπτωση όπου δεν ανανεώνεται ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνία σε ένα νεότερο. Πάντα να καλύπτουμε μια ε, παλαιά τέτοια περίπτωση. Δεν ξέρω αν αυτό γίνεται κατανοητό όλοι συμφωνούν ότι χρειαζόμαστε καινοτομία για τα φάρμακα και πρέπει να παράγονται όσο το δυνατόν φθηνότερα. Το σύστημα το οποίο λειτουργεί σήμερα δεν έχει και τα χειρότερα χαρακτηριστικά όσον αφορά αυτές τις δύο περιπτώσεις. 1,5% όσον αφορά την πραγματική έρευνα. Το ένα υπόλοιπο 15% αναπτύσσει με διαδικασίες στο φάρμακο και συγκρίνοντας τα στοιχεία από τη ΣΥΠΑ σε σχέση με ε, πάμπολα φάρμακα, 90% αναπτύχθηκαν με κονδύλια δημόσια όσον αφορά τη φαρμακοβιομηχανία. Είναι αυτό το πιο αποτελεσματικό σύστημα για να αναπτύσσουμε νέα φάρμακα και με αυτόν τον τρόπο παράγονται ή ε, έχουμε δυνατότητα να παράγουμε τα νέα αυτά φάρμακα με την μέγιστη επίπτωση στις αρρώστιες ή μήπως έχουμε ε, και θέμα όσον αφορά την προσιτή τιμή των φαρμακών. Διερωτώ με αν μπορεί το υφιστάμενο σύστημα να δώσει λύσεις ε, στα προβλήματα που έχουμε στην, ε, σήμερα και ακόμα και για την έκθεση που παραπονούνται όταν αρχίζει η έρευνα δεν γνωρίζουν ποια θα είναι η τελική έκβαση και στο δικό σας έγγραφο για τα την κάλυψη των δαπανών. Για τα αντιβιωτικά αυτό είναι κάτι πάρα πολύ λογικό, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις. Στις ε, μελέτες σας εξετάσατε το τι μπορεί να γίνει για να υπάρχει ενίσχυση στην έρευνα, γιατί διαφορετικά οποιοδήποτε μπορεί ένα γενώσιμο φάρμακο να το παράγει. Αυτό θα γινόταν και αυτό από πλευράς έκθεσής σας όταν το δίπλωμα ευρεσιτεχνία πάψει να ισχύει, αυξάνονται οι πωλήσει ενός φαρμάκου. Υπάρχει ζήτηση λοιπόν φαρμάκων και όμως ε, οι πολίτες δεν μπορούν να αγοράσουν κάποια φάρμακα επειδή είναι πολύ ακριβά και θα πρέπει να θέσουμε προτεραιότητες. Έχουμε φάρμακα λοιπόν που δεν είναι δυνατόν να είναι προσιτές οι τιμές διότι υπάρχει ε, το εμπόδιο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Ευρεσιτεχνίας έχετε εξετάσει εσείς το θέμα των τιμών. Δεν το είδα στις προτάσεις σας. Θα αποτελέσει τμήμα της αξιολόγησης οποιασδήποτε νέας μεθόδου. Προτού αρχίσουμε να έχουμε νομοθετήματα, νέες ε, νομοθετικές προτάσεις ε, για διπλώματα ευρεσιτεχνίας έχει μελετηθεί η βασική αρχή πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε να έχουμε αποτελεσματικά φάρμακα για τις ανάγκες μας. Well, κυρίως Γενικός. Μακάρι να μπορούσα και εγώ να το πω αυτό, ότι ο, η νομοθεσία για τον ανταγωνισμό δίνει όλες τις απαντήσεις και τις λύσεις. Το θέμα της καινοτομίας για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Και όπως είπα προηγούμενα, θα πρέπει να δούμε ότι θα πρέπει να είμαστε με αρκετή αυστηρότητα να επιβάλλουμε κανόνες σε αυτόν τον τομέα. Όμως παραμένει ένα πρόβλημα και αν παραμένει υπερβολικά μεγάλο πρόβλημα για την κοινωνία, για όλους μας αυτό, τότε αναπόφευκτο είναι ότι προβλήματα όσον αφορά τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας θα μεταφέρονται στα εσείς περιπτώσεις ανταγωνισμού. Για τον ίδιο τον ανταγωνισμό αυτό είδαμε από τις ΙΠΑ και είναι οι πρώτες που αναγνώρισαν αυτό το οποίο αναφέρθηκε πιο πριν, την ανάγκη προστασίας της καινοτομίας. Στην πρακτική εφαρμογή υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία εξελίσσονται και που δυστυχώς οδηγούν είτε σε αποδυναμωμένα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, είτε το αποτέλεσμα αυτών των ομάδων ευρεσιτεχνιών που σε σχέση με την, αντί να ενδυναμώσει την καινοτομία, την αποδυναμώνει. Επειδή δεν είναι απόλυτα σαφές πάντα ποια δικαιώματα είναι εκείνα τα οποία πρέπει να προστατεύονται και ποια είναι εκείνα τα οποία μπορούμε να εκμεταλλευόμαστε με τις ε, δέουσες διαδικασίες έβρεση τεχνίας. Έχετε λοιπόν δίκιο θα έλεγα ότι πρέπει να το τονίσουμε αυτό, ότι δεν είναι μόνο τα γενώσιμα που δημιουργούν προβλήματα όσον αφορά τα διπλώματα, τις ευρεσιτεχνίες, αλλά το σύνολο της βιομηχανίας χρειάζεται, της φαρμακοβιομηχανίας χρειάζεται ένα καλύτερο πλαίσιο για την καινοτομία και ένα καλύτερο πλαίσιο για τη διεξαγωγή του ανταγωνισμού. Και αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους ε, ε, έχουμε εμπλακεί συντάσσοντας και συστάσεις ε, δεν θα θέλαμε να προδικάσουμε το τι ε, πρόκειται να γίνει για τον πιο αποτελεσματικό τρόπο διοργάνωσης των ευρεσιτεχνιών. Πιστεύουμε ότι το κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας θα ήταν κάτι το αποτελεσματικό. Όσον αφορά τώρα τις ε, διαδικασίες για την αντιστάθμιση και αποζημίωση ή επανόρθωση Price funds θα μπορούσαν να, να είναι μια τέτοια ε, αντιστάθμιση μόνο που εμείς ε, επικεντρωθήκαμε στο να διακριβώσουμε ποιες ήταν οι απόψεις της φαρμακοβιομηχανίας πρώτα και μετά βλέποντας το τι γίνεται σε σχέση με ε, τα θέματα αυτά ξεκινήσαμε με κάποιες μελέτες όσον αφορά την ε, συμπεριφορά και το τι κάνουν διάφορες εταιρείες. Τώρα, σε σχέση με κάποιες φαρμακοβιομηχανίες, όταν έρχονται και λένε ότι δεν έγινε σκεμμένα κάτι τέτοιο, αλλά συμφωνήσαμε ότι θα μπορούσε να υπάρξει πρόβλημα εκτός αν υπάρξει αντισταθμιστική δράση και αν ε, μπορεί να λειτουργήσει η ιδέα του Price Fund θα ήταν μία από τις λύσεις που θα μπορούσε ίσως να είναι ενδεδειγμένη. Στο τέλος τέλος ο, στόχος ε, του, της νομοθεσίας ε, για τον ανταγωνισμό πολλές φορές πρέπει να βοηθά να γίνεται κάτι καλύτερο για τους καταναλωτές κοινωνικά φυσικά και μέσα στην ίδια τη διαδικασία του ανταγωνισμού αυτό. Αλλά να σας το πω αυτό δεν ε, εξετάσαμε όλες αυτές ε, τις ε, διαδικασίες, τις μελέτες. Βλέπουμε και εξετάζουμε τις πιθανές καταχρήσεις και υποβάλλουμε προτάσεις που διαβιβάζονται τους ε, συναδέλφους της ε, Γενικής Διεύθυνσης ε, ΣΤΑΝΚΟ βλέποντας αν αυτές οι προτάσεις για τις αλλαγές που προτείνονται είναι εφικτές και μπορούν να λειτουργήσουν μέσα σε ένα ρεαλιστικό χρονικό διάστημα ώστε να υπάρξει κάποιο θετικό αποτέλεσμα για τους ασθενείς και τα συστήματα υγείας. Αλλά ταυτόχρονα στο μεσοδιάστημα θα δώσουμε συνέχεια στην εξέταση αυτών των θεμάτων και αν υπάρχουν ε, σωστές λύσεις που μπορούν να προταθούν θα τις εξετάσουμε μέσα στο πλαίσιο της επίλυσης συγκεκριμένων προβλημάτων και τα συγκεκριμένα αποτελέσματα που μπορεί να έχουν στον ανταγωνισμό. Ευχαριστώ. Χατζημαρκάκης. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν ευχαριστώ πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το κοπιώδες ε, έργο. Δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά τον ρόλο των κρατών μελών. Τα κράτη-μέλη είναι αρμόδια για την τιμολόγηση και την διαμόρφωση των τιμών. Έχουν αυτό το δικαίωμα από πλευρά τους. Εγώ θα ευχόμουν να υπήρχε μια μεγάλη ευρωπαϊκή αγορά, αλλά όμως δυστυχώς έχουμε 27 διαφορετικές δομές όσον αφορά τις τιμές, την τιμολόγηση. Τεράστιες επιπτώσεις έχει αυτό, όχι μόνο για τις τιμές, αλλά και για το χρονικό σημείο πότε υπάρχει καινοτομία που εισέρχεται στην αγορά, με ποιους λόγους και με ποιες αφορμές καθυστερείται και τι γίνεται μετά στη συνέχεια ποιες επιπτώσεις υπάρχουν για να στεφτεί με επιτυχία. Ερώτησή μου, εσείς ως Επιτροπή μπορείτε να παροτρύνετε τα κράτη-μέλη την αποκαλούμενη οδηγία για την διαφάνεια, για την πολιτική τιμολόγηση να την χρησιμοποιούν και να τηρούν τις προθεσμίες, τις διορίες. Υπάρχει αυτή η διορία και προφανώς τα κράτη-μέλη δεν τηρούν τα υπεσχημένα μέσα στο πλαίσιο αυτό που είχαμε εμεί ω νομοθέτες ή συνομοθέτες σχεδιάσει. Ερώτηση, εσείς Ω Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση την ανάλυση τι κάνετε για να τηρούνται αυτέ οι διορίες. Αν αυτό το διασφαλίζαμε θα είχαμε κάνει ένα μεγάλο βήμα προ τα εμπρό. Η δεύτερη ερώτηση αφορά το evergreening, το πρασίνισμα. Είναι μία μέθοδο για να διευρύνεται το πλαίσιο μια τεχνία, ενό διπλώματο τεχνία. Έγιναν πολλέ συζητήσει και με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Τεχνιών και καταλήγουμε όλο και περισσότερο στο συμπέρασμα, και εγώ καταλήγω σε αυτό, ότι έχει νόημα αυτό όταν διευρύνουμε για μία περίοδο πέντε ετών ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, να το κάνουμε, αλλά μετά να υπάρχει μία αυστηρή τομή. Δηλαδή, άμεσα για το evergreening, αμέσως να το αναγνωρίζουμε και να το απαγορεύουμε. Μεγαλύτερο διάστημα προστασίας ευρεσιτεχνίας και μετά clear cut, σαφής παύση, λήξη. Ερώτησή μου, με αυτόν τον τομέα, όσον αφορά την ανάλυση σας, Πώς θα αντιμετωπίζατε αυτή την πρόταση, διότι πολλοί και από το γραφείο Ευρεσιτεχνίας του Μονάχου θεωρούν ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να ήταν κάτι το θελκτικό και θα είχε ωφέλη. Ευχαριστώ. Δύο αντιδράσεις. Ε, και δεν με καλύπτουν και 27 επιτροπή για αυτό που θα πω. Καταρχάς για την οδηγία διαφάνειας. Φυσικά, η Κομισιόν με μια έτσι στεναρή προσέγγιση θα μπορούσε να επικρίνει τα κράτη-μέλη, θα μπορούσε να τα απειλήσει με διαδικασίες επί παραβάση. Αλλά αυτό είναι όμως κάτι που δεν λειτουργεί απόλυτα, γιατί οι διαδικασίες αυτές είναι ε, χρονοβόρες οι αρχέ ανταγωνισμού στο εσωτερικό τη Κομισιόν έχει μπορούν να αντιδράσουν ε, στη... για μεγάλες εταιρείε στα κράτη-μέλη ή για εταιρείε που θεωρούμε ότι θα μπορούσαν να καταχρώνται δια... της κατάστασης θα μπορούσαμε να τις, να τις πιέσουμε αυτές τις εταιρείες ανεξάρτητα από την νομική πίεση. Ούτως ή άλλως αυτές οι εταιρείες ε, είναι οι πιο εκτεθειμένες για άμεση νομική αγωγή. Και το γεγονός ότι αυτές τις έρευνες τις κάναμε ε, ω σώμα από πλευρά Επιτροπή, ακριβώς ε, δίνουμε το σήμα ότι αυξάνουμε την πίεση για τις εταιρείε και τα κράτη-μέλη. Ένα δεύτερο, που είναι λίγο θεωρητικό. Αν ε, επιμηκύνουμε την ε, διάρκεια προστασίας, εν συνεχεία, ε, θα μπορούσαμε να πούμε τώρα stop. Εγώ νομίζω ότι, προσωπικά έτσι, ότι είναι ένας πολύ υγιής τρόπος να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα και προτιμώ αυτό παρά αυτές τις αχλαμάρες των συνεχών διαφορών ενώπιον δικαστηρίου και παρατάσεων κτλ. κτλ. Το πρόβλημα με αυτή την ιδέα είναι ότι ναι μεν είναι απλή, αλλά περιβάλλεται από δέσμε και συστάδες διπλωμάτων ευρεσιτεχνία. Ε, υπάρχουν συνάδελφοι στην Κομισιόν που έχουν μεγαλύτερη εμπειρία για αυτά τα θέματα. Εμείς απλώ είμαστε παρατηρητέ. Ε, εγώ θα έλεγα λοιπόν, ε, καλό θα ήταν να έχουμε κάτι σαφέ, απλό και να πούμε ότι τώρα, ας πούμε, ήρθε η στιγμή να σταματήσουν αυτές οι πρακτικές. Αλλά θα πρέπει να δούμε τα πράγματα κατά περίπτωση. Ευχαριστώ, κύριε Γενική. Ο κύριος ε, Παγνιέ. Όπως είπε... Όπως, πριν από λίγο ο πρέπει να σας αναγνωρίσουμε ότι ε, θέλησατε να προχωρήσετε σε αυτή τη θετική κίνηση αυτό το κειμένο τη ανακοίνωση και επίσης είναι πάρα πολύ θετικό το ότι έχετε αυτή την πρόθεση. Συνέχεια βλέπω ότι δεν προχωρήσατε όμως ε, με αρκετή τόλμη όσον αφορά αυτή τη διαδικασία την αντιμονοπολιακή ε, ε, του δικαίου του ανταγωνισμού γιατί αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα της δημόσιας υγείας θα το έχουν και οι Ευρωπαίοι της αύριο αυτό το επιστώνουμε όλη όλοι σήμερα και δυστυχώς θα το αντιμετωπίζουμε και στο μέλλον. Δεν έχω ερώτηση αυτή. Στον παρατήρησα το λέω. Και έχουμε όσον αφορά την ενημέρωση των ασθενών με έναν κανονισμό και μια οδηγία και όσον αφορά τις ε, διαφημίσεις των φαρμάκων θα πρέπει να αφήνουν περιθώριο τόσο ώστε να καλυφθεί το κείμενό σας και στη συνέχεια να τροποποιηθούν αντίστοιχα αυτά τα νομοθετήματα. Όμως δεν υπάρχει σωστή ισορροπία δυνάμεων όσον αφορά εμά και την άλλη μεριά τη φαρμακοβιομηχανία στην Ευρώπη. Θεωρώ, όπω και για την πολιτική ομάδα, ότι τα κράτη-μέλη σήμερα δεν έχουν τα απαραίτητη ισχύ ούτω ώστε να μπορέσουν να πιέσουν προ αυτή την κατεύθυνση τη φαρμακοβιομηχανία. Όντως, αυτό διαπιστώθηκε και στη Γαλλία σε σχέση με την γρήπη των χείρων και τα σχετικά εμβόλια και επίσης το θέμα είναι το τιμολογιακό όπως είπε και ο συνάδελφος για τα γενώσιμα. όπου υπήρχε πρόβλημα σε σχέση με τον των πωλήσεων. Ε, επομένως, θα πρέπει να προχωρήσουμε στη χαράξη μιας αυθεντικά κοινωνικής πολιτικής και να μην αφήνουμε τα κράτη μέλη να ενεργούν μια που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν επαρκώς της φαρμακοβιομηχανίας που είναι οργανωμένα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τρίτον, εκτός από το τιμολογιακό, σε σχέση με αυτή την ισορροπία δυνάμεων για την δημόσια υγεία, να δούμε πώς θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε καλύτερα τους καταναλωτές. Πρόσφατα εδώ συζητούσαμε και λέγαμε ότι στην Ευρώπη οι καταναλωτές δεν εμπιστεύονται τα φάρμακα. για να μπορέσουμε να χαράξουμε μια καλύτερη πολιτική, μια που δεν προκύπτουν λύσεις αναγκαστικά από τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Και να υπάρχει επιτέλους μια εμπιστοσύνη περισσότερο όσον αφορά τους φύλακες των συμφερόντων των κατάλληλων. Να υπάρχει επίσης μια πολιτική έρευνα και καινοτομία. Και αυτό να γίνεται, αυτή η πολιτική να ασκείται σε συνεργασία από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και να μην αφήνεται μόνο στα χέρια κάποιων επιχειρήσεων φαρμακευτικών. Βεβαίω και δεν μπορούμε να αφήσουμε στο παιχνίδι τι φαρμακοβιομηχανίε. Είναι ανάγκη αυτή η πολιτική έρευνα και καινοτομία. Και Εν κατακλείδη, νομίζω ότι με το κείμενό σας καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε κι άλλα. Ακόμα δεν υπάρχουν απαντήσει όλα τα ερωτήματα, αλλά θα πρέπει να λάβουμε τι ευθύνε μα και εμεί εδώ ως νομοθέτες ε, και χέρι με χέρι μαζί σας να μπορέσουμε να χαράξουμε μια πορεία με αναγκαία ισορροπία. Έχετε να μας πείτε δύο λόγια, ούτως ώστε να κλείσει η συζήτηση. Λόγω. Πρώτο πρώτο. Σε σχέση με εκείνους που θεωρούν ότι περιοριστήκαμε στα θέματα της τιμολογικής πολιτικής, αλλά όχι ε, στα γενικότερα, σφαιρικότερα προβλήματα του, του, κλάδου, πριν είναι αυτή η έρευνα είχαμε 27 υπουργούς. 27 κυβερνήσει. που θεωρούσαν στον τομέα της ενέργειας ότι υπάρχει μια εθνική ε, ενεργειακή πολιτική και ότι μπορούσαν να δημιουργήσουν κάποιες ευκαιρίε για την κοινωνία, για τους καταναλωτές γενικότερα. Όμως, είχαμε μόνο 10 εταιρείε στο σύνολο της Ευρώπης για το 99%, για το 95%, 95% της προσφοράς Βλέπετε επομένω ότι τεράστια ισορροπία υπάρχει μεταξύ αυτών που εκπροσωπούν τα συμφέροντα του συνόλου των Ευρωπαίων και των άλλων. Και βλέπετε επομένω τι είδου ισορροπία δυνάμεων και συσχετισμό δυνάμεων υπάρχει και που θα πρέπει επομένω αυτή η πορεία να διορθωθεί. Θα πρέπει να καταβληθεί επομένω αυτή η σχετική προσπάθεια και θα πρέπει αυτό να γίνει με την εφαρμογή του κανόνα του ανταγωνισμού. Και στο συγκεκριμένο σημείο συμφωνώ με το ότι θα πρέπει να βοηθήσουμε, να ενθαρρύνουμε την καινοτομία, την έρευνα και ανάπτυξη επίσης. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείε, κυρίως με αυτές που έχουν έδρα στην Ευρώπη. Και έχει δίκιο ο βουλευτής που είπε ότι δεν προχώρησε όσο θα έπρεπε, δεν ήμασταν στο έπρεπε με αυτή την έκθεση. Να κάτσουμε να δούμε τι, τι χρήματα το, το, το, το σύστημα προνοίας μας τόσα πολλά που θα πρέπει αντίστοιχα να προσέξουμε το πώς διαμορφώνονται οι τιμές και να δούμε ακριβώς και προσεκτικότερα τι σχέση υπάρχει μεταξύ των, ε, ε των, γενώσεων και των αρχαιοτύπων. Να κάτσουμε να δούμε τι χρειάζεται ο καταναλωτής, τι μπορεί να κάνει για να το βοηθήσει η αγορά. Σα ευχαριστώ και πάλι. Euh, Ευχαριστούμε κύριε Γενικέ, λέει πρόεδρο. Ευχαριστούμε για την εκθεσή σα τώρα κάπω ε, φωτίστηκε το τοπίο περισσότερο. Ε, Βεβαίω ακόμα κρυμούν πάρα πολλά ερωτήματα. Ε, αναπάντητα, ακριβώ όπως ε, είπαν οι, οι βουλευτές. Πάντω οπωσδήποτε είναι χρήσιμη η ενημέρωση που μα κάνατε και γι' αυτό και σα ευχαριστούμε ακόμη μια φορά εξ όλων. Euh, να συνεχίσουμε τις εργασίες μας, όχι με το θέμα της προστασίας των ακτών, που θα το εξετάσουμε στις 2 του μηνός, 2 Δεκεμβρίου, αλλά με το θέμα την πολιτική ποιότητας των γεωργικών προϊόντων. Πώς ε, θα μπορέσουμε να απλουστεύσουμε τη μελλοντική γεωργική πολιτική. Αυτό είναι το ερώτημα. Έχουμε μια έκθεση για αυτό το θέμα της κυρίας Πιλάρα Γιούζο. Αν θέλετε, κυρία μου, μπορείτε να μας παρουσιάσετε την έκθεσή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Αυτή είναι μια έκθεση της Επιτροπής που εστιάζεται σε θέματα που είναι σημαντικά για το μέλλον της γεωργικής πολιτικής και για το μέλλον προϊόντων ποιότητας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όπου πρέπει αυτό να το λάβουμε υπόψη. Η έκθεση αφορά κάποιες γεωγραφικές, γεωγραφικούς προορισμούς, ε, χαρακτηρισμούς ε, προέλευσης ε, και προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συγχωνευθούν τα δύο συστήματα των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ονομασιών. Και εγώ προσωπικά και η πλειοψηφία επίσης των μελών της Επιτροπής Γεωργίας είμαστε κατά αυτής της συγχώνευσης, διότι θα υποβαθμίζαμε τις ε, ε, ονομασίες προέλευση που έχουν τέτοια αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και η προστατευόμενη ονομασία προέλευση τουλάχιστον για το κρασί συνεπάγεται ότι παράγεται και επεξεργά, το εμφιαλώνουμε και το επεξεργαζόμαστε στον ίδιο τόπο της παραγωγής και θα ήμουν εναντίον να υπάρξει οποιαδήποτε αλλίωση του συστήματο να συγχωνευθούν δηλαδή αυτά τα δύο συστήματα με, γεωγραφικές, ε, με γεωγραφικούς προσδιορισμούς ε, όσον αφορά το σύστημα προσδιορισμού προστατευόμενων ονομασιών προϊόντων και όσον αφορά και την ε, αναφορά της ποιότητας και το χαρακτηρισμό ποιότητας, το μόνο προτέρημα θα ήταν μια διοικητική απλούστευση όπου το βάρος που αυτή τη στιγμή θα πρέπει να επομίζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες θα ήταν ελαφρότερο όσον αφορά τα πολλαπλά αιτήματα που υπάρχουν ε, για την ε, ρύθμιση των ε, προστατευόμενων ονομασιών. Υπάρχει όμως ο κίνδυνος να έχουμε πρώτης κατηγορίας και δεύτερης κατηγορίας προστατευόμενες ονομασίες και δεν θα έπρεπε να αλλάξουμε το υφιστάμενο σύστημα. Όχι μόνο να διατηρήσουμε το σύστημα αυτό, αλλά και να καθορίσουμε με καλύτερο τρόπο την, ε, τον ευδιάκριτο χαρακτήρα τους για τους Ευρωπαίους καταναλωτές, ώστε να υπάρχει πρόσθετη αξία όσον αφορά τα προϊόντα ποιότητας και όσον αφορά και τις γεωγραφικές, ε, τους γεωγραφικούς ε, χαρακτηρισμούς όσον αφορά την προέλευση όσον αφορά για το κρασί, για παράδειγμα και τα προϊόντα ποιότητας, πιστεύω ότι θα πρέπει να παραμείνει το σύστημα ως έχει. Το ε, σύστημα για το κρασί που ε, ήταν παλαιότερο και μετά υπήρξε ο επιπροσδιορισμός των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης. Πιστεύω ότι αν υπάρξει συγχώνευση θα υπάρξει σύγχυση όσον αφορά την ε, αναφορά προέλευσης όσον αφορά εκείνους που θα εμπλέκονται στην διαδικασία αυτή. Στο διεθνές πλαίσιο θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να βελτιωθεί να βελτιωθεί η προστασία των δικών μας ονομασιών προέλευσης προϊόντων από πλευρά της Ευρώπης και που έναντι προϊόντων απομίμησης πρέπει να είμαστε αυστηροί για να τα προστατεύουμε τα προϊόντα μας, ιδιαίτερα τα κρασιά. Και όσον αφορά την ε, εμπορία, ο καθορισμός των πρώτων υλών όσον αφορά την γεωργία βελτιώνει σίγουρα σε σχέση με την μεταποίηση προϊόντων. Όμως υπάρχει το πρόβλημα βάρος που μπορεί να δημιουργηθεί, της επιβάρυνσης ε, που δεν νομίζω ότι ε, θα ήταν ε, δικαιολογημένη. Η αναφορά δηλαδή σε σχέση με τις πρώτες ύλες για τα μεταποιημένα προϊόντα θα πρέπει με βάση, σε θελοντική βάση να μπορεί να γίνεται σε σχέση με το να αποφύγουμε υπερβολική επιβάρυνση όσον αφορά τους όσους θα εμπλέκονται σε αυτό το σύστημα για την ε, αναφορά της προέλευσης ε, αυτών των ε, ουσιών. Και σε σχέση με την ενιαία οριζόντια ρύθμιση με εγκάσιο χαρακτήρα όλων των κανόνων που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε ένα, ας το κάθετο πλαίσιο και έχοντας υπόψη την ρύθμιση που υπάρχει αυτή τη στιγμή αν αλλοιώναμε αυτό το πλαίσιο θα αφήναμε στα χέρια ιδιωτών την διατήρηση και διαχείριση των ονομασιών. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τις ονομασίες που αυτή τη στιγμή υφίστανται διασφαλίζοντας με μια, μια μεγαλύτερη διαφάνεια για την αγορά όσον αφορά αυτά τα προϊόντα και η δική μου στάση, η δική μου θέση είναι να διατηρηθούν αυτές οι προδιαγραφές για την προστασία των προϊόντων και δεν θα ήθελα να αφήσουμε να αναλάβουν οι ιδιώτες την ε, ε, διαχείριση αυτού του πλαισίου. Είμαι όμως θετική για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για νέες, ε, νέους προσδιορισμούς που για παράδειγμα θα μπορούσε σε εθελοντική βάση να λειτουργεί με, όσον αφορά την ορεινή γεωργία και τις καλλιέργειες καθώς επίσης ε, και όσον αφορά τις ε, ε, εκπομπές ρήπων διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό θα πρέπει να το αφήσουμε για μια ιστερότερη φάση όσον αφορά την ρύθμιση αυτού του θέματος του διοξιδίου του άνθρακα. Και όσον αφορά τα νέα συστήματα πιστοποίησης, μελετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την εισαγωγή ε, ετικετοποίησης όσον αφορά ε, τη ζωική προέλευση ε, ή την προέλευση των τροφίμων όμως θα πρέπει εδώ να δούμε ότι πρόκειται για μια επιβάρυνση για την θέσπιση ενός ευρωπαϊκού καθεστώτος ρύθμισης. Πρέπει να υπάρξει μια γενική καταχώρηση κοινοτική συνολικά. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να μπορεί να γίνεται μια εκστρατεία προώθησης ε, των προϊόντων αυτών και αυτού του είδους της γεωργίας, διότι στο τέλος τέλος είναι στοιχεία αξιόλογα για τον καταναλωτή αυτά. Και όσον αφορά την οικολογική ετικέτα που υφίσταται, είμαι θετικά διακείμενη στο να υπάρξει ένα νέο λογότυπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την ε, ε, προώθηση αυτών των προϊόντων στην αγορά. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλές διαφορετικές ετικέτες, ε, οικολογικές και άλλες. Έχουμε 17 διαφορετικά τέτοια, διαφορετικές τέτοιες ετικέτες στη χώρα μου και αυτό δημιουργεί σύγχυση στον καταναλωτή. Και όσον αφορά τις, ε, τη ρύθμιση για την ε, κρατική πιστοποίηση, συμμερίζομαι απόλυτα την πρόταση για το τι θα μπορούσε αυτό να συνεπάγεται στην ενιαία ε, αγορά και να υπάρχει η δυνατότητα αυτή να ρυθμίζεται με ενιαίο τρόπο. Είναι αναγκαίο λοιπόν να υπάρξουν μέτρα ώστε στο μέτρο του εφικτού να υπάρξουν ε, ενιαίες ετικέτες ε, ποιότητας που θα αναγνωρίζονται μέσα από ένα πλαίσιο αμοιβαίας αναγνώρισης. Και έτσι αυτό θα είναι ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός αν το καταφέρουμε. Στο τέλος θα ήθελα να πω σε την προώθηση των προϊόντων ποιότητας ότι σε αυτή την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πολύ μεγάλη σημασία η προαγωγή των προϊόντων ποιότητας όχι μόνο όσον αφορά το κρασί και όπως γίνεται και με την κοινή οργάνωση αγοράς για τον Ίνο, αλλά και όσον αφορά την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μεγάλο μέρος του προϋπολογισμού για την ε, προώθηση και προαγωγή του ε, κρασιού όσον αφορά τρίτες ε, χώρες αντιμετωπίζει προβλήματα. Είναι αναγκαίο λοιπόν να έχουμε ένα ενιαίο πλαίσιο για την προαγωγή αυτών των προϊόντων μέσα και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Euh, Ευχαριστώ κύριε Συγγήτρια για τη θαυμάσια εισαγωγή σας. Ο κύριος Μάριο Πυρίλο έχει το λόγο, αν το επιθυμεί. Αγαπητή Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον την έκθεση της εισηγήτριας. Φυσικά το θέμα είναι πολύ παλιό. Οι ονομασίε των γεωργικών μας προϊόντων εγώ προέρχομαι από μια έντονα γεωργικά περιοχή, όπου έχουμε συζητήσει πάρα πολύ την αναγνώριση των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων. Και συμφωνώ απόλυτα με την εισηγήτρια ότι πρέπει να διατηρήσουμε τη διάκριση για να μην ε, δημιουργήσουμε σύγχυση μια τόσο δύσκολη χρονική στιγμή για τη γεωργία και για τα γεωργικά προϊόντα της Ευρώπης. Κάτι άλλο θα ήθελα να πω τώρα για τα βιολογικά γεωργικά προϊόντα. Τα βιολογικά προϊόντα, έχετε δίκιο αγαπητοί συνάδελφε, μπαίνουν στην αγορά με διάφορα λογότυπα. Στη χώρα σας έχουμε 17 διαφορετικά λογότυπα. Φανταστείτε τι γίνεται σε επίπεδο 27 κρατών μελών. Νομίζω ότι για αυτό το θέμα θα πρέπει να δώσουμε κι εμείς μια άποψη. Πιστεύω ότι με ένα ενιαίο σήμα, με ένα ενιαίο λογότυπο, θα δώσουμε μια σωστή απάντηση σε αυτούς που σήμερα προτιμούν τα βιολογικά προϊόντα. Τα βιολογικά προϊόντα, μην ξεχνάτε ότι έχουν τεράστια επιτυχία. Και στη δική μου χώρα, στην Ιταλία και στην περιοχή μου, τα βιολογικά προϊόντα ε, έχουν μεγάλη απήχηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρώση. Ευχαριστώ. Και εγώ άκουσα με προσοχή τις παρεμβάσεις των προηγούμενων ομιλητών και ιδίως της εισηγήτριας και συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με αυτά τα οποία είπε. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το να διατηρήσουμε χωριστές της ονομασίας προέλευσης από τις γεωγραφικές ενδείξεις, γιατί πραγματικά θα μπορούσε να δημιουργηθεί σύγχυση αν τις ανακατέβαμε στο μυαλό του καταναλωτή. Έχω μία ανησυχία, μία αμφιβολία για ένα πολύ σημαντικό θέμα. Δηλαδή, τι πρέπει να έχει τελικά η ετικέτα. Γιατί ενώ από τη μία σε πολλά προϊόντα είναι αδύνατο να χρησιμοποιήσουμε τον όρο ευρωπαϊκό προϊόντο, ε, προϊόν, συγγνώμη, γιατί για να έχουμε ένα ευρωπαϊκό τελικό προϊόν θα πρέπει να έχουμε και ευρωπαϊκές πρωτεσίλες, αλλά σε αυτή την περίπτωση έρχονται από άλλες χώρες. Επομένως θα, μπορούσαμε να πούμε στην ετικέτα ότι κάποια τμήματα του προϊόντος δεν προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αυτό ε, δημιουργεί πρόβλημα στην επιχείρηση που θέλει να πουλήσει το προϊόν. Αυτό είναι το ένα. Από την άλλη όμως είναι άσχημο να βγάλουμε κάποιες ονομασίες από την ετικέτα ή να μην προβλέπουμε τέτοια δυνατότητα. Γιατί? Ε, με αυτόν τον τρόπο δεν αξιολογούμε, δεν προωθούμε προϊόντα τα οποία ε, παράγονται από πρώτες ύλε που προέρχονται από ξένες χώρες. Ε, είναι άσχημο όταν σέβονται βέβαια τις, ε, τα, τα πρότυπά μας, καλό να τα προωθήσουμε. Αλλά υπάρχει περίπτωση να προέρχονται από προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούν, ας πούμε, εντομοκτώνα, ε, ζυζανιοκτώνα. Ε, εμείς τα απαγορεύουμε. Σε άλλες χώρες όμως επιτρέπονται. Επομένως δεν πρέπει να τα προωθούμε αυτά τα προϊόντα. Ε, το τελικό προϊόν, το οποίο στο εσωτερικό του περιλαμβάνει τέτοιες ουσίες απαγορευμένες, ε, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στον καταναλωτή. Το να μην το βάλουμε στην ετικέτα σημαίνει ότι δεν δίνουμε ενδείξεις ε, στον ε, καταναλωτή. Ένα παράδειγμα του μελιού. Που, ένα θέμα που το συζητούσα με έναν Ιταλό συνάδελφο, που είναι ένα κλασικό Ιταλικό προϊόν. Υπάρχουν ε, εταιρείε που λένε ότι το μέλι το οποίο αγοράζεται είναι ε, εξωτερικής προέλευσης. Ε, δεν προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. άλλοι δεν το λένε ή άλλοι το λένε, ότι παράγεται στην Ιταλία στη συγκεκριμένη ε, περιοχή. Το να μην βάλουμε αυτές τις ενδείξεις ε, σημαίνει ότι βάζουμε ε, μέσα στο, στο κουτί, ας πούμε, μέλι κατώτατης ποιότητας και το πουλάμε, λες και παράγεται στην Ιταλία, χωρίς καμία διάκριση. Αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Αυτό που ρωτάω λοιπόν τους συναδέλφους και κυρίως την εισηγήτρια είναι να προσέξουμε πάρα πολύ για να δούμε πώς μπορούμε να συγχωνεύσουμε τις δύο απαιτήσει. Δηλαδή, να έχουμε ευδιάκριτες ετικέτες για το καταναλωτή, ε, κατανοητές, αναγνώσιμες, από την άλλη να εξασφαλίσουμε όμως και την παροχή της πληροφορίας ε, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος ε, η κυρία. κυρία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την κυρία Γιούσο για την εκθεσή της και επειδή έκανε αυτή την εισαγωγή από πλευρά της. Πρέπει να έχουμε το θέμα αυτό μπροστά μας και να συνειδητοποιούμε περί τίνος πρόκειται για την πολιτική, για την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων και ποια στρατηγική πρέπει να ακολουθήσουμε η κυρία Γιούσο πολύ σωστά αναφέρθηκε στην προέλευση, γεωγραφική προέλευση και χαρακτηρισμό γεωγραφικό των προϊόντων αυτών που είναι ένα χαρακτηριστικό ποιότητας για αυτά. Αυτό το χαρακτηριστικό ποιότητας κάπως κλειδονίζεται σε αυτή την περίοδο. Διότι ο ένας στρέφεται κατά του άλλου ή έχουμε ανταγωνισμό και ανταγωνιζόμαστε μεταξύ μας. Και τώρα στόχος μας πρέπει να είναι να βρούμε μια λύση που να είναι στραμμένη προς το μέλλον, που θα μας συνενώνει όλους σε ένα ενιαίο πλαίσιο. Και έχουμε κοινέ αρχές και βάσεις. Αυτές οι κοινέ αρχές καθορίζονται και κατοχυρώνονται σε αυτό το κείμενο στην ε, οργάνωση αγοράς της ευρωπαϊκής πολιτικής ε, για αυτά τα προϊόντα. Και γι' αυτό θα πρέπει κοινό παρανομαστή και κοινά στοιχεία ως Ευρωπαίοι να αναζητήσουμε ως ένα σύμβολο ή λογότυπο για τις διαφημίσεις για τέτοιου είδους προϊόντα και την οικονομική πτυχή και το ποιοτικό χαρακτηριστικό αυτών των προϊόντων που πρέπει να αναφέρουμε που έχει παραχθεί σύμφωνα με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σύμφωνα με την cross-compliance, την συνολική συμμόρφωση για τις ε, αρχές της γεωργικής πολιτικής. Διότι αυτή η cross-compliance διασφαλίζει μια αηφορία στην παραγωγή και πρέπει εδώ, θα έλεγα, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος να είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για μας. Η αηφορία στην παραγωγή, η αηφόρος παραγωγή τροφίμων με υψηλή ποιότητα ποιοτικών τροφίμων παραγωγή και επιπλέον αηφορία όσον αφορά το τοπίο, το περιβάλλον μας, διατήρηση και προστασία των τοπίων και της υπαίθρου. Να δώσουμε ιδιαίτερο βάρος σε αυτά τα στοιχεία. Και αυτά έχω υπόψη όταν λέω ότι σε ένα παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο οικονομίας θα είναι δύσκολο η καθαρή αρχή προέλευσης του προϊόντος να καθορίζεται 100%. Ας πάρουμε την πίτσα για παράδειγμα. Να λέμε μόνο από την Ιταλία. Ε, δημιουργούνται ήδη προβλήματα όσον αφορά τις διάφορες ουσίες, ως συστατικά αυτής της πίτσας, που ίσως δεν είναι όλες οι Ιταλικές ένα χαρακτηριστικό ποιότητας πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο επικέντρωσης για μας και να πούμε είναι μια ονομασία ιταλική για αυτό το προϊόν και μιας περιφέρειας ίσως, αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι υποχρεωτικό, γι' αυτό υποστηρίζω την εθελοντική προσέγγιση, εθελούσια βάση που προτείνει η κυρία Αγιούσο για το χαρακτηρισμό ποιότητας και προέλευσης και αηφορία όσον αφορά τα τρόφιμα και τη γεωργική, την παραγωγή <laughs> αυτών των τροφίμων από τη γεωργία και για όλα τα γεωργικά ευρωπαϊκά προϊόντα αυτό πρέπει να είναι η αρχή και στο τέλος είναι σημαντικό να καθορίζονται αυτά έτσι στην αγορά και έτσι με αυτά τα στοιχεία με τους όρους και προϋποθέσεις πώς θέλουμε να παράγονται αυτά τα στοιχεία θα μπορούσαν να είναι χαρακτηριστικά ποιότητας για αυτά τα προϊόντα. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ κυρία Κλάς. κύριος Ρίχτερ. Ένα σχόλιο σύντομα. Και αυτό είναι ότι συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι εδώ δεν πρέπει να αποδυναμωθούν οι χαρακτηρισμοί ποιότητα όσον αφορά την προστασία, προστατευόμενη ονομασία προέλευση ή συγκεκριμένου ε, χαρακτηρισμού και χαρακτηριστικά όσον αφορά προστατευόμενα προϊόντα. Δεν πρέπει να αποδυναμώσουμε αυτέ τι αρχέ, Αλλά υπάρχει και η ετικέτα τη χώρα προέλευση. Και μία από τι πιο συχνέ ερωτήσει είναι από πού προέρχεται το τρόφιμο αυτό, το φαΐ αυτό. Όταν αγοράζει κανεί για παράδειγμα μια πίτσα, άσχετα αν έχει παραχθεί στην Ιταλία ή στην Γερμανία, από πού προέρχεται το κρέας που χρησιμοποιείται στην παραγωγή μιας πίτσας. Αυτό θέλουν οι καταναλωτές να γνωρίζουν. Οι καταναλωτές που θέλουν να αποφεύγουν μεγάλες οδούς, μεγάλες αποστάσεις στις μεταφορές, έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν από πού προέρχεται ένα προϊόν και οι συστατικές του ουσίες. Γιατί οι συστάσεις αυτές το βρίσκω θετικό. Η Επιτροπή Γεωργίας το Μάρτιο είχε καθορίσει με σαφή τρόπο μια σαφή διάταξη και ένα σαφές πλαίσιο για την, ε, τον καθορισμό της προέλευσης. Αναχώρα. Εγώ θα το χαιρέτιζα αν μπορούσαμε αυτό να το προχωρήσουμε πιο πέρα ακόμα και να το μεταξελίξουμε. Αυτό θα το συζητήσουμε και όσον αφορά την ετικετοποίηση και τη συσκευασία στο μέλλον. Όμως συμφωνώ απόλυτα με την Επιτροπή Γεωργίας που θεώρησε ότι ο προσδιορισμός της προέλευσης είναι ένα μέσο, ένα εργαλείο για τους καταναλωτές για να μπορούν να επιλέγουν το προϊόν που επιθυμούν σύμφωνα με τις αρχές που επιθυμούν. Πρέπει να το διατηρήσουμε ώστε να μην υπάρχει οποιαδήποτε σύγκρουση με τις γεωγραφικές ονομασίες προέλευσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ προσθέτω την άποψή μου και συμφωνώ με την εισηγήτρια. Θεωρώ και εγώ την σκόπιμο αυτά τα δύο συστήματα να διατηρηθούν ως έχουν, διότι έχουν λειτουργήσει σωστά ακριβώς για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη Γεωργία είναι τεράστια σημασία ε, να μπορούν ε, με αυτές ε, τις βάσεις να συνεχίσουν να διοχετεύουν τα προϊόντα τους στην αγορά. Και δεν επιτυγχάνει η συγχώνευση αυτών των δύο μέτρων και συστημάτων δεν επιτυγχάνει αυτό που θέλουμε. Να καθίσταται σαφές για τους καταναλωτές ότι για κάποια προϊόντα, για κάποια τρόφιμα η αναφορά για τα, τη γεωργική, την ε, γεωγραφική προέλευση του προϊόντος ή την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης που είναι πρόθυμοι οι καταναλωτές να πληρώσουν και κάτι παραπάνω για να αγοράσουν ένα τέτοιο προϊόν και όσον αφορά την... Ε, δεν πρόκειται για το ότι το ένα είναι καλύτερο από το άλλο ή το άλλο ή μπορεί να είναι χειρότερο, αλλά υπάρχει η πρόθεση όταν γνωρίζουν οι καταναλωτές ότι μια συγκεκριμένη διαδικασία έχει γίνει σεβαστή και έχει χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ενός προϊόντος, να πληρώσουν κάτι παραπάνω ως τιμή. Και τώρα συνολικά <clears throat> όσον αφορά είχαμε και μια, την έκθεση ε, υποσυζήτηση, πρέπει να προσέξουμε να μην υπάρξουν υπερβολικές επιβαρύνσεις και διαφορές και εναλλακτικέ δυνατότητες όσον αφορά τα τρόφιμα. Θα δημιουργηθεί σύγχυση και δεν θα υπάρχει μια συνοπτική εικόνα για το ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος. Καμιά φορά λοιπόν ένα μικρότερο πλαίσιο μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικό από ένα ευρύτερο και πιο ε, λεπτομερές ε, ε, σύστημα. Εδώ επίσης ε, θα πρέπει να έχουμε και την δυνατότητα να μπορούμε μέσω φορέων πιστοποίησης ε, να αντιμετωπίσουμε την ανεξέλεγκτη τάση κάποιων ιδιωτών ε, να πιστοποιούν τα δικά τους προϊόντα και να αναφέρουν ότι έχουν παραχθεί με τον ένα ή άλλο τρόπο. Εδώ λοιπόν με θετικό τρόπο, επικοδομητικό πνεύμα πρέπει να υποβληθούν τέτοιες προτάσεις στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ζέμπερ. Κύριε Ντελάνγκ παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να πω ότι εδώ θα πρέπει, αντιδρώντας ε, σε σχέση με τον κύριο Σλούτερ, ο Ολλανδός καταναλωτής θέλει να ξέρει ποιο τυρί βρίσκεται στην πίτσα και αν είναι πραγματικό τυρί, ή αν είναι υποκατάστατο τυριού. Το κάθε κράτος, η κάθε, ο κάθε πολίτης, ανάλογα με τη χώρα από την οποία προέρχεται, έχει τις δικές του προτιμήσεις ε, και τις δικές του συνήθειες. Ε. Και εφόσον λοιπόν όταν υπάρχει μια διαφοροποίηση μεταξύ δύο κατηγοριών, όταν έχουμε τον πρωτογενή προϊόν ε, τομέα και όταν έχουμε ε, και την μεταποίηση, είναι πολύ σημαντικό με βάση τα όσα είπε η κυρία Κλάς. Οι απαιτήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι πολύ υψηλότερε από εκείνε ε, που αντιμετωπίζουν κάποιοι οι ιδιώτες σε πιο περιορισμένο πλαίσιο. Αυτό πρέπει να το δούμε. Και την εθελοντική βάση ε, χαρακτηρισμού από, σε σχέση με τη χώρα προέλευσης ή την γεωγραφική, τον γεωγραφικό προσδιορισμό ενός προϊόντος. Εντάξει, με εθελοντική βάση να γίνεται αυτό όπως λέει η κυρία Γιούσο. Όμως εθελοντική χρήση αυτών των επισημάνσεων δεν θα πρέπει να οδηγεί σε σύγχυση και ούτε θα πρέπει να είναι εμπόδιο στην ελευθερία κυκλοφορίας και διακίνησης. Όσον αφορά την, ε, το, το λογότυπο, το σύμβολο της ε, βιολογικής γεωργίας ε, θα έπρεπε ήδη να υπήρχε πανευρωπαϊκά. Αλλά δεν υπάρχει ακόμα, διότι έχουμε κάτι το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά και στο λογότυπο Aldi και αυτό έχει δημιουργεί, προβλήματα. Όμως το ευρωπαϊκό λογότυπο θα πρέπει οπωσδήποτε να μπορέσει να τεθεί. Μάλλον κιόλα εξεπλάγει ότι ήταν ε, η Επιτροπή Προπολογισμών πρόθυμη να, να, να διαθέσει περισσότερα κονδύλια όσον αφορά ε, την δυνατότητα ελέγχου των ε, εισαγόμενων προϊόντων να δουν αν ανταποκρίνονται σε σχέση με τις προδιαγραφές όπως θα έπρεπε. Όμως δεν διατέθηκαν κονδύλια για αυτούς τους ελέγχους τελικά. Και όσον αφορά τις εκπομπές ε, ρήπων, διοξιδίου του άνθρακα, ίσως εδώ ε, ένας ορισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα ε, ήταν αναγκαίος διότι διαφορετικά η κάθε υπεραγορά, σούπερ μάρκετ, στο, η Τέσκο για παράδειγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει ένα λογότυπο χαμηλής ε, επιβάρυνσης του περιβάλλοντος με διοξίδιο του άνθρακα σε σχέση με τις ε, διαφορετικές ε, δυνατότητες προσδιορισμού οι διαφορετικούς ορισμούς που υφίστανται. Οι διαφορές είναι τόσο μεγάλες που χάνει πια νόημα να έχουμε διαφορετικά λογότυπα για αυτά τα προϊόντα πρέπει να έχουμε ένα ενιαίο λογότυπο. Αυτά ήθελα να πω. Είναι μια εξαιρετική έκθεση η έκθεση της κυρίας Αγιούσο. Ε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Πριν σα ξαναδώσω το λόγο, κυρία εισηγήτρια, να δώσω το λόγο σε κάποιον που ξέχασα προηγουμένω. Έχετε το λόγο. Σα ακούμε. Μικρόφωνο σας παρακαλώ. Μικρόφωνο παρακαλώ. Το μικρόφωνο σας δεν λειτουργούσε. Ευχαριστώ. Ε, αυτό που ήθελα να τονίσω σε μια έκθεση που φαίνεται να είναι ενδιαφέρουσα είναι ότι καλούμαστε να ορίσουμε μια πολιτική ποιότητα των γεωργικών προϊόντων ε, και τη στρατηγική της μέσα σε ένα ανταγωνιστικό διεθνές πλαίσιο ε, και σε ένα περιβάλλον όπου η κοινή αγροτική πολιτική για μας πρέπει να πάρει υπόψη της και αυτό το πλαίσιο και με δεδομένο ότι ε, ακολουθείται μια πολιτική μείωση των ε, αγροτικών δραστηριοτήτων και του πληθυσμού των αγροτών και οι οποίοι προφανώς πρέπει να δουν ταυτόχρονα και πολιτικές προστασίας του εισοδήματός τους. Ε, η μόνη διέξοδος ε, σε αυτό το διεθνές πλαίσιο και αρνητικό για τους αγρότες ε, κυρίως της Νότιας Ευρώπης. Η μόνη διέξοδος λοιπόν είναι τα ποιοτικά προϊόντα. Αυτά είναι προφανώς και τα προϊόντα ονομασίας προέλευσης και τα βιολογικά, τα οποία και πρέπει να εξασφαλιστεί για τα οποία πρέπει να εξασφαλιστούν η έλεγχοι και η πιστοποίηση ώστε να προστατεύεται και ο καταναλωτής αλλά και τα συμφέροντα αυτών οι οποίοι κάνουν πραγματική δουλειά και σέβονται και τον καταναλωτή. Ε, εμείς υποστηρίζουμε και ταυτόχρονα με την προστασία του περιβάλλοντος και της αισθητικής και την υγεία των ανθρώπων και των οικοσυστημάτων, αλλά θα θέλαμε και την ενίσχυση των συλλογικών μορφών παραγωγής, την ενίσχυση των ομάδων παραγωγής, ή ακόμη ε, την, ε, κάτι που είναι πολύ σημαντικό, την ε, αποφασιστική πολιτική κατά της εισβολής και διάδοσης των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Αποτελεί χαρακτηριστικό σημείο ε, υπεράσπισης της ποιοτικής παραγωγής. Επιπλέον, η ενίσχυση της τοπικής παραγωγής έχει να κάνει τελικά, ε, εκτός παραγωγης εχει να κανει τελικα εκτος απο την προστασία του εισοδήματος, και με την προστασία του πλανήτη. Και θα πρέπει να συνδυάζεται με πολιτικές αποθάρρυνσης των ε, μεταφορών. Διότι μπορεί ένα προϊόν να ε, παράγεται σε κάποια μακρινή περιοχή με βιολογικό τρόπο, αλλά δεν είναι ποιοτικό και οικολογικό τελικά, ακριβώς γιατί στην εποχή της κλιματικής αλλαγής θα πρέπει να παίρνουμε σοβαρά υπόψη ότι ε, επιβαρύνει τον πλανήτη με τα καυσαέρια τα οποία ε, εξοδεύονται για να έρθει στον Ευρωπαίο καταναλωτή. Με αυτή την έννοια η εξασφάλιση ποιοτικών ε, προϊόντων έχει να κάνει και με τις αντίστοιχες πολιτικές στις ε, μεταφορές και την προστασία του περιβάλλοντος. Θα θέλαμε λοιπόν αυτή η τοπική παραγωγή, οι συλλογικές μορφές και ποιοτικές βιολογικές θα λέγαμε εμείς μορφές παραγωγής θα πρέπει να ενισχύονται και μέσα από εκθέσεις σαν και αυτή που θα πρέπει να, ε, και να την προστατεύσει και μέσα από συγκεκριμένες πρακτικές μορφές όπως ε, είναι τα λογότυπα, οι έλεγχοι, οι πιστοποιήσεις αλλά και η ένταξη αυτής της πολιτικής σε αυτό το γενικό πλαίσιο στο οποίο αναφέρθηκα. Αν δεν υπάρχουν άλλοι που να θέλουν να πάρουν το λόγο, η κυρία εισηγήτρια. Αλλά θα ήθελα και εγώ να σας θέσω μια ερώτηση που σας δώσω το λόγο για να απαντήσετε. Στο σημείο 12 προτείνεται να ενθαρρύνουμε την ολοκληρωμένη παραγωγή, όπως λέτε. Δεν φοβάστε ότι θα δημιουργηθεί μια επιπλέον σύγχυση, αν λάβουμε υπόψη όλα όσα είπαμε ε, για τις ε, επισημάνσεις βιολογικών προϊόντων. Εγώ συμφωνώ να αφήσουμε τα δύο συστήματα, γεωγραφικές ενδείξεις και ονομασίες προέλευσης δηλαδή. Και συμφωνώ ότι πρέπει να αναπτύξουμε μια γεωργία που να προστατεύει το περιβάλλον και να προωθεί και τα βιολογικά προϊόντα. Αλλά αυτή η ολοκληρωμένη παραγωγή. Τι νόημα έχει, μια και οι κανόνες που έχουμε λάβει είναι ούτως ή άλλως πολύ αυστηροί σε ό,τι αφορά ειδικά τα ζυζανιοκτώνα. Τα φυτοφάρμακα γενικά. Ε, αυτά μπορείτε να απαντήσετε τώρα και σας ευχαριστώ για την ποιότητα της έκθεσης. Ευχαριστώ και θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους παρενέβησαν για τις παρεμβάσεις τους και τα σχόλιά τους θα πω όσον αφορά την ολοκληρωμένη παραγωγή στη συνέχεια μέσα στο πλαίσιο της ενιαίας ε, γεωργικής πολιτικής υπάρχει μια, ε, ένας μια ρύθμιση για την παραγωγή τροφίμων ε, το καλύτερο θα ήταν όμως ε, από αυτή την έκθεση να μην το ε, εντάξουμε σε αυτό, διότι αναφέρεται αυτή η έκθεση στην πρόσθετη αξία και τις προδιαγραφές ε, παραγωγής πρόσθετης αξίας όσον αφορά την αναβάθμιση και σε σχέση με την χρήση συγκεκριμένων προϊόντων. Επιπλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν προπομπή, ήταν πρωτοπόροι για αυτές τις ε, διαδικασίες παραγωγής ε, όπως ε, και για την ονομασία προστατε... γεωγραφική προστατευόμενη ονομασία και χαρακτηρισμούς γεωγραφικής προέλευσης. Πρέπει να συνεχίσουμε διατηρώντας αυτές τις επισημάσεις και πέρα από την οικολογική βιολογική γεωργία και εκείνο που θέλω να πω είναι να υπάρξει ένα λογότυπο ευρωπαϊκό και να μην εμπέσουμε στην, ας το έτσι, ε, φρούδα ή μη καρποφόρα ε, λύση στο να έχουμε εκατοντάδες, ε, δεκάδες διαφορετικά τέτοια λογότυπα όσον αφορά την ρύθμιση της οικολογικής γεωργίας και των προϊόντων της. Ένα ενιαίο λογότυπο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και η ρύθμιση, η προστασία όσον αφορά την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης και τους χαρακτηρισμούς αυτών των προϊόντων που είναι μία, ας το πω έτσι, ε, προδιαγραφή ε, διασφάλισης παραγωγής ε, προϊόντων και για την γεωγραφική, ας πούμε, τον γεωγραφικό καθορισμό επιπρόσθετα. Έχοντας αυτό το σύστημα, για παράδειγμα, όσον αφορά το αμπέλι, το σταφύλι, για την παραγωγή και την αμπελοκαλλιέργεια σε ένα συγκεκριμένο σημείο, για παράδειγμα στον Μπορντό, για την γεωγραφική αναφορά. Αυτό σημαίνει ότι μπόρεσε να παραχθεί ένα ε, από το αμπέλιτο ε, στα όμως ε, μέσα στο πλαίσιο μιας ε, γεωγραφικής περιφέρειας, μέσα στο σύστημα αυτό της ε, ε, ονομασίας, ε, γεωγραφικής ονομασίας, ο Ευρωπαίος καταναλωτής έχει συνηθίσει να αναγνωρίζει και γνωρίζει τα προϊόντα αυτά. Θα έχουμε μεγάλη σύγχυση που θα δημιουργήσουμε αν αυτά τα συστήματα τα αλλοιώσουμε και πάψουν να ισχύουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ την εισηγήτρια για τη θαυμάσια προσπάθειά της. Υπενθυμίζω ότι η ημερομηνία για την κατάθεση των τροπολογιών είναι 8 Δεκεμβρίου στις 12 θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή ΕΝΔΗ 25 ε, με 27 Ιανουαρίου 2010 στην Επιτροπή ε, Άγκρη Φεβρουάριο 2010 και στην Ολομέλεια το Μάρτιο του 2010. Ε, σταματάω εδώ τη συνεδρίαση μέχρι αύριο το πρωί. Ήμασταν αρκετά σύντομοι σήμερα. Αύριο το πρωί λοιπόν θα τα πούμε. Γεια σας. Mm.